Okay, colleagues. Συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης είναι η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση πάνω στη Συμφωνία TTIP. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση σήμερα το πρωί και ξέρω πως οι συνάδελφοι σκιώδες γιατί εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά για να καταλήξουμε σε αυτούς τους συμβιβασμούς. Ελπίζω λοιπόν η ψηφοφορία να είναι εύκολη. Χθες όταν άρχισε η συνεδρίαση είχαμε αναβάλει την ψηφοφορία για τα ορυκτά που αποτελούν αντικείμενο συγκρούσεων για το Στρασβούργο. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν για αυτό σήμερα, αλλά το Μάρτιο, στις 9 Μαρτίου. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά πρώτα ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, αν είμαστε εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία. Ας πούμε, ποιος θέλει να πιει τσάι, ψηφίστε. Οι σοσιαλιστές <laughs> θέλουν, βλέπω. Κάτι διαδικαστικό, είναι Δεν έχω την κάρτα μου, θα σας δείξω με το χέρι λοιπόν. Okay, I think in that case you can... Μάλιστα, μπορούμε να σας συνυπολογίσουμε λοιπόν. Οι υπόλοιποι έχετε τις κάρτες σας. Ωραία. Okay, well people are just coming in. It's working. Βλέπω έρχονται και άλλοι, το σύστημα λειτουργεί. Πέρας. Ωραία, η πλειοψηφία θέλει να πιει τσάι. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Κα... Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Πρόσθετη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Στη σελίδα 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 28. Και αυτή προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 καταπίπτει. Τροπολογία 41. Προσθήκη και αυτή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Τώρα πάμε στη σελίδα 7, τροπολογία 43. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 ως προσθήκη είναι στη σελίδα 8. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 προσθήκη υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 68 και 69 είναι ταυτόσιμες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 10 ως προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 στην σελίδα 11, έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σαρλ ε, Γκέρντς, προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82. Ψηφίσαμε το κείμενο με την προφορική τροπολογία και όχι την ίδια. Η προφορική τροπολογία έχει την προσθήκη το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Είναι ένα κείμενο δηλαδή που βρίσκεται εντός της προφορικής τροπολογίας. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μισό λεπτό. Πρόκειψε κάτι τεχνικής φύσεως. Μας λείπει κάτι Λυπάμαι συνάδελφοι, έγινε ένα λάθος και πρέπει να επιστρέψουμε στην τροπολογία 75 στη σελίδα 10. Τη βρήκατε? Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη Θέλω να στήσω, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε αυτή, για αυτή που ξεχάσαμε. 75, τη βρήκατε. Στα δικά μου ε, χαρτιά είναι στη σελίδα 10, σε άλλους μπορεί να είναι στη σελίδα 9. 75, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκαέξι ψήφοι υπέρ, επτά κατά, μία αποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Λίτς και όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή τους δουλειά. Καταφέραμε να έχουμε μία ομαλή ψηφοφορία. Ωραία συνάδελφοι, πρέπει να περάσουμε γρήγορα στο επόμενο σημείο γιατί δεν θέλουμε να αργήσει πολύ η ακρόασή μας, δεν θέλουμε να την καθυστερήσουμε. Παρακαλώ πολύ συνάδελφοι καθίστε και όλοι εσείς που έχετε πηγαδάκια εδώ και εκεί με στην αίθουσα τα πηγαδάκια εκτός εθούσης. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση ε, τώρα, ε, η οποία ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κάναμε καθυστερήσαμε τις ψηφοφορίες έτσι ώστε να έχουμε χρόνο όλοι και η ίντα μάλιστα καθυστέρησε την ψηφοφορία της θα την κάνει την 9η Μαρτίου έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ε, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα των ορυκτών σε ε, ζώνες ε, που βρίσκονται σε σύραξη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της κοινή γνώμης για το θέμα αυτό και εγώ λαμβάνω ηλεκτρονικό ταχυδραμείο. Take meetings outside. Το ξαναλέω λοιπόν, παρακαλώ πολύ, ησυχία, ηρεμία, όσοι θέλουν να συζητήσουν να πάνε εκτός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος έτσι ώστε να, μπορέσω, να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ε, το λόγο. Γιατί το θέμα, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην τελευταία συνεδρίαση του Στρασβούργου είχαμε ε, και άλλη μία συνάντηση ε, με τους σκιώδης για το θέμα αυτό τον Μάρτιο θα κάνουμε μία συνεδρίαση έκτακτη για να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είναι πολλές τροπολογίες, 200 μάλιστα. Ε, τις έχουμε τώρα στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Και ε, πρέπει να πω ότι εγώ τώρα προσπαθώ ε, μαζί με την ε, με την ομάδα μου να, κάνω, να, να δω τις τροπολογίες αυτές. Έχουμε προχωρήσει, βρισκόμαστε ήδη σε καλό σημείο. Η βάση λοιπόν της, ε, του συμβιβασμού ε, αντιπροσωπεύεται, βασίζεται στις τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Κυρίως τροπολογίες που έχει υποβάλει η ομάδα ALDE που επιθυμεί συμβιβασμό όπως και εγώ άλλωστε. Εγώ προσπαθώ να βρω έναν κοινό τόπο, κοινέ βάσεις όσον αφορά ε, τις διάφορες πολιτικές ομάδες, γιατί υπάρχει κοινό τόπος κατά την άποψή μου ε, και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο σε πολλά σημεία όπως είναι οι ζώνες ε, σύραξης, όπως είναι τα, οι πρώτες τα κτλ. Ναι, ε, νομίζω ότι ε, σημαντικό είναι να δούμε ποιες είναι οι απόψεις των μεν και των δε όσον αφορά τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να στείλουμε ένα σημαντικό, ένα καθαρό μήνυμα ε, μέσω της γνωμοδότησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια εγκάρσια συμφωνία, ε, συμβιβαστική ε, λύση μεταξύ των πολιτικών ομάδων και ελπίζω ότι η πλειοψηφία θα μπορέσει να επικυρώσει την, τις συμβιβαστικές προτάσεις. Θα έχω την δυνατότητα, ελπίζω και στο σύντομα, να μιλήσω με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρόμπερτ Νόιζερ ε, για τους σοσιαλιστές. Ε, μιλώ εκ μέρους ε, του Σεμπάστεν Ερτς, ο οποίος έχει τώρα την ίδια στιγμή μια σημαντική ψηφοφορία στην άλλη του Επιτροπή. Οι περισσότεροι πλέον είχαμε την δυνατότητα να κοιτάξουμε τις τροπολογίες ε, τροπολογίες οι οποίες έχουν ε, υπογραφεί από πολλούς ε, βουλευτές πολλών ομάδων. Είναι σαφές πλέον ότι πρέπει να αναλυφθεί δράση και είναι σημαντικό να υπάρξουν κοινοί τόποι. Ε, οι τροπολογίες αποτελούν ε, το, το αποτέλεσμα μιας ε, πολύμηνης προσπάθειας των, από πλευράς των πολιτικών ομάδων, από πλευράς των σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, το θέμα μας απασχολεί πολύ ε, και προσπαθήσαμε να ε, εμπνευστούμε από την αντίστοιχη αμερικανική νομοθεσία έτσι ώστε να και, να λάβουμε υπόψη μας και τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων. Θα πρέπει οι μηχανισμοί να είναι καλοί και για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες παίζουν κάποιο ρόλο σε όλη την αλυσίδα ε, της εκμετάλλευσης και της αλυσίδας εφοθιασμού. Οι τροπολογίες μας αντικατοπτρίζουν αυτό που πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη λύση έτσι ώστε ε, να σταματήσουν τα φαινόμενα ε, των, της προσπάθειας επιρροής ε, και ε, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να, ε, για να μπορέσουν να δουλέψουν χωρίς να υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις των σειράξεων. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, στα σύνορα της ε, Ευρώπης να υπάρχουν τέτοια άλυτα ζητήματα τα οποία, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα επιβίωσης ακόμα σε ανθρώπους που ζουν έξω από την Ευρώπη. θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του μέχρι ε, και το τέλος της ε, ε, αλυσίδας έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια πραγματικά σωστή απάντηση στα προβλήματα. Τα υπάρχοντα σχήματα δεν έχουν λειτουργήσει. Τώρα θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερες, ε, σε ακόμα περισσότερα σημεία σύγκλησης ε, θα πρέπει να ε, στηρίξουμε την ανάπτυξη και θα πρέπει να δείξουμε και τη διάθεση συνεργασίας που έχουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ο Λουί Μισελ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί πιστεύω ότι η προσέγγιση που έχει επιλέξει είναι σωστή. Είναι ε, ταυτόχρονα φιλόδοξη αλλά και λογική. Υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ουσιώδους ε, σημασίας αυτό που ανέφερε προηγουμένως δηλαδή ε, να μην γίνεται εθελοντική αυτοπιστοποίηση αλλά να υπάρχει ε, χαρακτήρας υποχρεωτικός. Πιστεύω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια καλή ευκαιρία ε, να, πάρει δράση, ε, να αναλάβει δράσεις έτσι ώστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου να γίνουν σεβαστά υπέρ της ειρήνης και της ευημερία. Εγώ ζητώ λοιπόν ενδυνάμωση του κανονισμού αυτού που θα έχει οπωσδήποτε ε, δεσμευτικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Είμαι αρκετά ε, υπέρ επίσης να υπάρξει ιδέουσα επιμέλεια σε όλη την αλυσίδα ε, εφοδιασμού γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν, ε, ελοχεύει μάλλον ο κίνδυνος να υπάρξουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί ένα ευέλικτο σύστημα ηχνηλασιμότητας και λογοδοσίας. Όσον αφορά δε τις υποχρεώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν και κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ε, ε, με το βάρος των επιχειρήσεων. Οπωσδήποτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία από ότι οι πολύ μεγάλες ε, ε, ε, επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε τον, την χάρτα του ΩΣΑ όσον αφορά αυτού του είδους της επιχειρήσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να οργανωθεί μια τέτοια παρακολούθηση έτσι ώστε όλη αυτή η ολοκληρωμένη διαδικασία να γίνεται βάσει καλών μεταρρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο. Ε, γιατί διαφορετικά, εάν δεν ακολουθήσουν με την απαραίτητη ε, διαρθρωτική προσαρμογή αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες έχουν ε, τέτοιου είδους ορυκτό πλούτο, τότε οπωσδήποτε οι συμφωνίε θα είναι μειωμένη σημασίας και οπωσδήποτε μειωμένη γεωγραφικής επάρκεια. Θα πρέπει οπωσδήποτε η προσέγγιση να είναι ε, ε, ολιστική ε, θα πρέπει να παρουσιαστούν οπωσδήποτε όπως έλεγα και προηγουμένως και τα απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα τα οποία εάν δεν υπάρχουν θα αποδυναμώνεται πάρα πολύ η πρόταση. Επίσης πιστεύω ότι ελοχεύει και κάποιος κίνδυνος ε, εάν δεν βάλουμε και έστω ένα χαμηλό επίπεδο κυρώσεων. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε διατυπώσεις όπως τα κράτη ενδεχομένως θα προσέξουν κτλ. Πρέπει να έχουμε ένα ε, έστω ελάχιστο επίπεδο ε, κυρώσεων. Ε, επίσης, ο καθορισμός των εμπολέμων ε, περιοχών ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει τις αρχές του οδηγού του ΟΣΑ. Θα πρέπει φυσικά να ζητούνται από τις, να υπάρξει διαβούλευση με τις επιχειρήσεις έτσι ώστε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε και τη θέση των εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, ε, πιστεύω ότι μια χρονική περίοδος δύο ετών είναι λογική ε, έτσι ώστε να επιτρέπεται και η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ενδιαφερόμενους γενικά αλλά και η δυνατότητα αναθεώρησης. Τέλος, καθορίζοντας σαφείς κανόνες που θα συνοδεύουν έναν σαφώς λειτουργούντα μηχανισμό, θα μπορέσουμε και να προστατέψουμε τις ντόπιε περιοχές, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επενδύσεων, αλλά και την ανάπτυξη των χωρών. Πιστεύω ότι ε, θα μπορέσουμε ε, να βρούμε μια πλειοψηφική συμφωνία όσον αφορά το θέμα αυτό. Thank you. Um, Κυρία Σαρζεντίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βασικό για μένα είναι αυτή η Επιτροπή, που είναι Επιτροπή Ανάπτυξης, να αποδείξει πως δεσμεύεται υπέρ του περιορισμού της χρηματοδότησης των σειράξεων που χρηματοδοτούνται από μεταλλεύματα και ορυκτά. Φοβάμαι ότι η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι υπερβολικά ευρωεμπορική. Εμείς πολλές φορές έχουμε πάει πιο μακριά, κάνοντας κάποιες νομοθετικές προσπάθειες που δεν πέτυχαν και νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες προοδευτικές προσεγγίσεις και να ξεκαθαρίσουμε με την ίντα πως το θέμα αυτό δεν είναι μόνο εισαγωγικό μέτρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και αναπτυξιακό εργαλείο για την ε, αποφυγή ε, σειράξεων. Για τους συμβιβασμούς λοιπόν του εισηγητή νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατανοεί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται πολύ στον κανονισμό του ΟΣΑ για την δέουσα επιμέλεια για την αλυσίδα νεφοδιασμού Και στις κατευθυντήριες γραμμές για τη δέουσα επιμέλεια του ΟΣΑ είναι ένας χαλαρός νόμος. Δεν είναι ένα σχήμα το οποίο απαγορεύει τις εισαγωγές και δεν είναι ένα καθεστώς το οποίο Χρειάζεται απλώς να συνδεύεται από ένα επιπλέον χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. δέουσα επιμέλεια προσπαθεί απλώς να πείσει όλους να κάνουν το σωστό και να βελτιώσει συντοχρόνω κάποια πράγματα. Φαίνεται λοιπόν πως Αυτό το ξεχνάμε και η μένη είναι υπέρ μιας υποχρεωτικής νομοθεσίας και ε, υπέρ μιας νομοθετικής ε, προσπάθειας ε, δέουσας επιμέλειας. Δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε τη χαλαρή νομοθεσία και γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ της ε, ε, επιμέλειας, της δέουσας επιμέλειας. Ε, είπε ο εισηγητής, άκουσα από τη Διερμηνία, ότι δεν είναι υπέρ της υποχρεωτικής νομοθεσίας. Α, δεν συμφωνούμε πια. Εγώ πίστευα ότι ήσασταν υπέρ προτάσεων που καταστούν αυτές τις αδειοδοτήσεις υποχρεωτικές. Thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλοι συνάδελφοι να ζητάνε το λόγο. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Κομισιόν, μάλιστα. Δεν έχω τα ονόματά σας, δεν ξέρω από πού είσαστε. Μάλιστα, είστε από την Γενική Διεύθυνση Trade και DevCo. Εντάξει, θα πάρετε και εσείς το λόγο. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τα σχόλια του Λουί Μισελ και των προτάσεων που κάνει για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω πως υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να συμπεριλάβουμε όλη την αλυσίδα του ε, φοδιασμού και να πούμε μόνο τα χιτήρια. Μη συγχωρείτε μόνο τις εγκαταστάσεις τήξης, γιατί στην ε, κατευθυντήρια γραμμή όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να, στην ε, κατευθυντήρια γραμμή για τη δέουσα επιμέλεια πρέπει να συμπεριλάμβονται όλες οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα όσα λέω όσα. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν την δέουσα επιμέλεια αλλά δεν καλύπτουν όλη την αλυσίδα της, ε, τον εφοδιασμό. Άρα λοιπόν ήθελα να σχολιάσει η Κομισιόν το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο ΩΣΑ. γιατί όταν το πρώτο συζητήσαμε είπαμε Έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ που ουσιαστικά λειτουργούν από το εφαρμόζεται του 2007. Πείτε μου λοιπόν, πόσες, ε, πόσες επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μεταλλεύματα σύραξης. Το 40%? Δεν θυμάμαι τι είχατε πει είναι, επαναλαμβάνω, μια εθελοντική ε, διαδικασία συμμόρφωσης και νομίζω γι' αυτό τώρα προχωράμε προς μια δεσμευτική ε, βέβαια εσείς είπατε εθελοντική αλλά για όλη την αλυσίδα νεφοδιασμού έτσι δεν είναι όχι μόνο για κάποια τμήματα πείτε μας λοιπόν κομισιόν και μετά ε, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να απαντήσει την κυρία Σαρτζεντίνη Αφού έχουμε λοιπόν εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α τα πει το δυνατόν πιο γρήγορα. σα παρακαλώ μην μακρηγορήσετε γιατί ο Επίτροπο σας περιμένει έξω να μπει. Για να απαντήσω στο θέμα που θέσατε, δεν έχω πολλά να προσθέσω σε σχέση με τα σχόλια των πολιτικών ομάδων. Να σας πω μόνο πως για την κατευθυντήρια γραμμή του ΩΣΑ και γιατί θεωρούμε πως αποτελεί βελτίωση με μεγάλη προστιθέμενη αξία προς τον κανονισμό, Σημαίνει τα εξή. Καταρχήν έχουμε ένα σύστημα επιβολή μέσω των ε, αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε το σύστημα αυτό του ΟΣΑ ή το σύστημα του κανονισμού, έτσι κι αλλιώ θα έχετε υποχρεωτικού ελέγχους και ε, αρμόδιες αρχές από τα κράτη-μέλη που θα επιβεβαιώνουν πώς ακολουθείτε αυτή την δέωση επιμέλεια. Δεν είναι ότι απλώς θα το δηλώνετε. Δεύτερον, έχουμε ε, έχουμε και ένα κατάλογο με χιτήρια και μεταλλουργία και νομίζω ότι αυτό καλύπτει και τη διάσταση της διαφάνειας που έχετε ζητήσει. Εμείς ε, απαιτούμε ελέγχους από τρίτα μέρη όχι μόνο για τα χιτήρια και τα μεταλλουργία όπως κάνει κατευθυντήρια γραμμή αλλά και για τους εισαγωγείς. Και αυτό επιπλέον με τα συνοδευτικά μέτρα τα οποία είναι κομμάτι της ε, σφαιρικής προσέγγισης που ακολουθούμε και φαίνεται στην ανακοίνωση της είπα ε, προσώπου. Είναι νομίζω αρκετό το σύστημα αυτό για να εξασφαλίσει στην αγορά πως έχουμε διαφάνεια, πως οι επιχειρήσεις ε, που είναι υπεύθυνοι εισαγωγής αναγνωρίζονται και πως αρκετές επιχειρήσεις ε, ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Γιατί η ισορροπία μεταξύ, του, μεταξύ κόστους και ωφέλους στην περίπτωση αυτή είναι σημαντική. Γιατί αποφεύγοντας τα αρνητικά αποτελέσματα μιας υποχρεωτικής, ενός υποχρεωτικού συστήματος και στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια και να καλύψουμε τις βασικές πηγές ανεφοδιασμού. Συνάδελφε, έχετε κάποια τελευταία σχόλια? Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε και να πατήσω πρώτα στην κυρία Σαρζεντίνη. Σε πολλές, ε, με πολλές ε, φωνές έχει απαντηθεί το ερώτημά σας. Και θα σας παραπέμψω στα εξή λεγόμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο και να ε, προχωρήσει στην εφαρμογή ενός υποχρεωτικού μηχανισμού. Ε, αυτή είναι η θέση μου, υποχρεωτικού. Κύριε Μισελ, η διαφάνεια είναι σημαντική. Παράλληλα όμως, πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα αυτό το οποίο θα χτίσουμε να εφαρμοστεί. Δεν αποκλείω να έχουμε και κάποια νομοθεσία κατάντη, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό συστατικό, αλλά σημαντικότερο ακόμα είναι να εξασφαλίσουμε προς τα πλαίσια του σχεδίου συμβιβασμού που θα σας ε, μοιράσω πριν τα τέλη της εβδομάδας θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και σε ποιο επίπεδο της αλυσίδας θα ε, τοποθετήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Ε, το υποχρεωτικό σύστημα πάντα ήταν η προτιμητέα λύση για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το απάντησες λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω και περιμένουμε να μας μοιράσετε αυτό το συμβιβασμό μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και ευχαριστώ όλους σας για τη σκληρή δουλειά που κάνετε έτσι ώστε να έχουμε μια μεγάλη επιτυχία. Κλείνω αυτή τη συνεδρίαση. Η επόμενη είναι 9 Μαρτίου του, στο Στρασβούργο. Δεν γνωρίζουμε την ώρα, αλλά έχει επιβεβαιωθεί γύρω στις 7 ή 7.30 σε 9 Μαρτίου. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα ψηφίσουμε... Α, συγγνώμη, στις 9.30 το βράδυ τη Δευτέρα, όχι 7.30, 9 Μαρτίου. 9.30 το βράδυ θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. 21 και 30. Δευτέρα, 9 Μαρτίου, επαναλαμβάνει η πρόεδρος. Άρα λοιπόν, παρακαλώ να φάτε πριν έρθετε. Και εκείνη τη στιγμή θα ψηφίσουμε για τα ορεκτά σειράξεων. Εγώ νόμιζα τα ψηφίσουμε σε 7.30. Μου είπαν τώρα στις 9.30. Στις 9.30 το βράδυ σημειώστε το τώρα στην ατζέντα σας. Να είστε εκεί. Είναι σημαντική η ψηφοφορία και σας χρειαζόμαστε όλους. Και επόμενη συνεδρίαση 31 Μαρτίου, 3 ε, το απόγευμα και 9 το πρωί, 1η Απριλίου. Κλείνει λοιπόν η συνάντηση της Επιτροπής μας και περνάμε στην ακρόαση. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τον κύριο Περέιρα να ανέβει στο πόντιο. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, έτσι ώστε να αρχίσουμε αυτή την ακρόαση για τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να κάνουμε αυτή την ακρόαση. Έχουμε διακεκριμένους πανελίστες και όπως ξέρετε αυτό το θέμα θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής το επόμενο έτος. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για την ε, αναπτυξιακή χρηματοδότηση και ο εισηγητής, κύριος Περέιρα, θα είναι πρόεδρος στην σημερινή ακρόαση, μάλιστα. Θα γίνει διάσκεψη στην Αντίσα τον Ιούλιο και ξέρουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει κάποιες προτάσεις για την χρηματοδότηση ανάπτυξης. Τους επόμενους μήνες θα προετοιμάσουμε την έκθεσή μας. Ο κύριος Πέντρος Σίλβα Περέιρα είναι ο εισηγητής και καλέσαμε εσάς για να μας εκθέσετε τις απόψεις σας για το ζήτημα αυτό, πώς μπορούμε να κάνουμε πρόοδο, πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία στη Νέα Υόρκη. Χωρίς καθυστέρηση όμως θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή κύριο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Λίντα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σήμερα το απόγευμα στην ακρόασή μας για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης δηλαδή. Σήμερα θα συζητήσουμε για το πώς θα επιτύχουμε τους, ε, αναπτυξιακούς, ε, τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Έχουμε διακεκριμένους καλεσμένους σε δύο πάνελ. Στο πρώτο πάνελ θα πάρει πρώτο το λόγο ο Επίτροπος Μίμητσα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις παρουσίασε τις δικέ της προτάσεις με μορφή ανακοίνωσης. Ανυπομονούμε λοιπόν να ακούσουμε τα σχόλιά σας για την ανακοίνωση αυτή. Επίσης, Έχουμε μαζί μας τον Jesse Griffith, τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Χρέος και την Ανάπτυξη, το Eurodad, το οποίο δίκτυο έχει ηγετικό ρόλο στην αναπτυξιακή χρηματοδότηση και συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικές με την ανάπτυξη. Επίσης, και εμεί, η δική μα Επιτροπή, προετοιμάζει τη δική τη ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σίγουροι πώ θα μα βοηθήσετε σε αυτό το έργο. Επίσης, θα μου ο Chris West, ο οποίο είναι διευθυντή του Ιδρύματο Shell και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ε, Αναπτυξιακού Ινστιτούτου με μακρόχρονη πείρα σε θέματα ανάπτυξης. Με χαρά μας λοιπόν θα ακούσουμε και τη δική σας προοπτική, την επιχειρηματική προοπτική στην αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Έπειτα, στο δεύτερο πάνελ, να σας πω ότι δυστυχώς δεν θα είναι πλήρως το πάνελ, διότι ο Υπουργός που είχαμε καλεσμένο από την Αιθιοπία δεν κατάφερε να έρθει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θα έχουμε λοιπόν καλεσμένους. Την Γκέιλ Χέρλι που είναι πυρογνώμονα στο... στα πλαίσια της διάσκεψης των Ηνωμένων Αθηνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Και τον James Jean Διευθυντή του Τμήματος ε, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων της, ε, του Τμήματος των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη. Είμαστε εδώ κυρίως για να ακούσουμε τους καλεσμένους μας. Λίγα σχόλια θα χωρέσουν. Φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη είναι η σημασία της διάσκεψης στην Αντισαμπέμπα διότι θα δώσει τον τόνο για τις επόμενες διασκέψεις στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο για τους ε, στόχους αηφορίας στην ανάπτυξη και αργότερα το Δεκέμβριο στη διάσκεψη για το κλίμα. Όλοι φυσικά εμείς στηρίζουμε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα έτσι ώστε να δημιουργηθούν ισχυρές παγκόσμιες συνεργασίες για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και φυσικά όλοι συμμεριζόμαστε τις απόψεις για τον ε, καταμερισμό της ευθύνης. Όλοι έχουμε ευθύνη Ιδιαίτερα δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι χώρες τις ίδιες δυνατότητες. Ιδιαίτερα μετά από τις ε, εξελίξεις των τελευταίων ετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετικό ρόλο στην όλη διαδικασία Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καλωσορίζουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει δείξει μια πολιτική δέσμευση για την ανάπτυξη καθώς και πολιτική συνοχή έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Έχει έρθει η ώρα όμως να αρχίσουμε την ακρόση. Ήδη υπόθηκαν κάποια πράγματα σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής και ελπίζουμε σήμερα το απόγευμα να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, μιλώντας για τις επίσημες δεσμεύσεις στα πλαίσια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει και να επιβεβαιώσει τους ε, δεσμευτικούς στόχους του 0,7%. Και το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την συμφωνία που θα γίνει στη διάσκεψη της Αντισαμπέμπα. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν σήμερα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ ο Πίτροπος Μίμητσα και θα ακούσει τις απόψεις μας και εμείς τις ε, δικές του. Είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει αυτός ο στόχος για το 0,7% του καθαριστού εθνικού εισοδήματος σε αναπτυξιακή βοήθεια, όμως αυτός ο στόχος πρέπει να γίνει και πραγματικότητα και πρέπει να κερδίσουμε αξιοπιστία. Και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλοι φορείς στους στόχους αυτούς. Δεν θα σταθούμε όμως μόνο στο θέμα της ε, αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Θα συζητηθούν και οι εγχώροι πόροι, διεθνή συστήματα φορολόγησης, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και πώς θα, θα συμπεριληφθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στους ε, στόχους μας. Δεν θα καθυστερήσω όμως άλλο. αλλά θα δώσω το λόγο αμέσως στον Επίτροπο Μίμητσα, ευχαριστώντας τον ξανά για την παρουσία του εδώ μαζί μας σήμερα. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διαστόματος Επιτρόπου, καθώς και τις πρώτες αντιδράσεις τις οποίες έχουμε ήδη πληροφορηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Σιγητά, αγαπητέ Πέδρο. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, αυτή η ακρόαση έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη ε, καμπή όσον αφορά την ε, διαπραγμάτευση για την ατζέντα μετά το 2015, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο πιο θερμό του σημείο στην ε, Νέα Υόρκη. Σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών υπάρχει μεγάλη εστίαση στο θέμα αυτό. καταφέραμε αρκετά. Ε, έχουν προταθεί από το Open Working Group 17 στόχοι οι οποίοι ε, αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο μέρος ε, του, τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως καταγράφτηκαν στην ανακοίνωση του Ιουνίου του 2015. Αυτή τη στιγμή η εστίαση μετατίθεται στον τρόπο πώς δηλαδή θα οργανώσουμε τη δράση μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να υλοποιήσουμε αυτήν ε, την φιλόδοξη ατζέντα, αυτό το θεματολόγιο το οποίο ε, προχωράει, ε, πηγαίνει από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την επιστηστική βοήθεια και τις πρώτες ύλες, περνώντας από μια σειρά άλλα στοιχεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε σώσουμε τον πλανήτη και τη ζωή των ανθρώπων. Το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σας τον προηγούμενο Νοέμβριο καλούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση των νέων ε, συνολικών εταιρικών σχέσεων που είναι απαραίτητες μετά το 2015. Και στα συμπεράσματα του 2014 ε, ε, καλείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί. Εμείς ανταποκριθήκαμε Βρεθήκαμε λοιπόν στις εκκλήσεις σας ε, και ε, στις 100 μέρες της νέας Κομισιόν συμπεριλάβαμε και το θέμα αυτό ε, που δείχνει πόσο μεγάλη σημασία το αποδίδουμε. Στην ανακοίνωση της 15ης Φεβρουαρίου λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, αναφέρεται ότι η Global Partnership είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση αυτού του θεματολογίου. Βασιζόμαστε σε αρχές όπως είναι η καθολικότητα και η επιμερισμένη ευθύνη. Ε, υπογραμμίζουμε επίσης την ανακοίνωση αυτή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, την ισότητα των φύλων, ε, την έλλειψη διακρίσεων κτλ. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια, έναν κατάλογο σωστών του to-do list, για όλες τις χώρες. Στην ανακοίνωση επίσης αναφέρονται συγκεκριμένες και πλήρες προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος, επιθεώρηση και λογοδοσία. Στη, θέλουμε η ανακοίνωση αυτή να αποτελέσει βάση ε, για, την, ε, για τον μελλοντικό γεφυρωτικό και επικοδομητικό ρόλο που θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ σε τρία στοιχεία ιδιαίτερα τα οποία πιστεύω ότι βρίσκονται, έχουν ένα ε, μια πυρηνική σημασία και που μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα συζήτησης σήμερα. Η συνολικότητα λοιπόν είναι ένα σημαντικό ε, θέμα το οποίο θίγεται στην ε, ε, ανακοίνωσή μας. Δεν είναι δυνατόν οι ενέργειες που θα γίνουν να είναι μεμονωμένες. Οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να είναι συνολική και όχι μεμονωμένη. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει, να, θα η χρηματοδότηση αυτή να παίξει καταλητικό ρόλο κυρίως στις χώρες οι οποίες περισσότερο χρειάζονται την χρηματοδότηση αυτή. Θα πρέπει όμως να το βάλουμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Επομένως, η ανακοίνωσή μας υπογραμμίζει επίσης και την ε, ε, σημασία του να μην υπάρχουν ODA ε, πολιτικές επιλογές. η δυνατότητα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ε, η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης, ε, η δυνατότητα, ε, η δυνατότητα δημιουργίας γηγενών πόρων, εγχωρίων πόρων, μέσα και από τις δυνατότητες φορολόγησης, μέσα και από τις ενδεχόμενες ε, την ενδεχόμενη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία μπορούν να ε, ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να, έχει, που μπορεί να έχουν οι σωστές διαδικασίες παρακολούθησης, επιθεώρησης και λογοδοσίας θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία ενδυνάμωση, αμοιβαία επιλογή αλλά και συμπληρωματικότητα ε, τώρα ακόμα περισσότερο από πριν έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε το Σεπτέμβριο σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι λογικό, σωστό, συνολικό και συνεκτικό και το οποίο να μπορέσει να αποτελέσει βάση για κοινωνική και περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. για, την, ε, ε, για το θεματολόγιο μετά το 2015 θα πρέπει να δούμε ε, όλες τις δυνατότητες, εγχώριες και αλλοδαπές, κοινωνικές και εμπορικές. Θα πρέπει να δούμε μια νέα ατζέντα για το 2015 και μετά. Το δεύτερο σημείο είναι η καθολικότητα, universality ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική ε, εσωτερικά και εξωτερικά. Θα πρέπει να υπάρξει από το 2015 και μετά μία μετατόπιση ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση όλων των χωρών. Δεν είναι δυνατόν πλέον να ακολουθήσουμε την επιλογή της συνηθισμένης εργασίας. Το business as usual δεν μπορεί πλέον να ισχύει πιστεύω ότι μέσω της ανακοίνωσής μας ε, μπαίνουμε πλέον επικεφαλής αυτού του μετόπου και είμαστε πλήρως διατεθειμένοι να παίξουμε το ρόλο μας και όχι μόνο να ενθαρρύνουμε και άλλους να παίξουν το δικό τους ρόλο. Η δημόσια ε, παγκόσμια χρηματοδότηση θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο για αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλά έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τις δηλώσεις της χιλιετίας του 2000. Βαθμιαία αυξήσαμε την χρηματοδότησή μας έτσι ώστε να φτάσουμε στο 0,73% του ΑΕΠ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, 75 δις ευρώ περίπου. Αυτό είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο του ΩΣΑ και ε, αντιπροσωπεύει τεράστια αύξηση παρά τις ε, μεγάλες ε, οικονομικές δυσκολίες, πολύ μακριά από το 0,32% που είχαμε μερικά χρόνια πριν. Ε, πάνω από περίπου το μισό της παγκόσμιας βοήθειας ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρότι η ίδια περνάει μέσα από δυσκολίες οικονομικές. Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα ε, πολύ χαμηλά όσον αφορά ε, την πορεία προόδου για την πλήρη επίτευξη του στόχου, ωστόσο πολλά έχουν γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να φτάσει τον στόχο του 0,7%. Επίσης πιστεύουμε ότι και οι περιφερειακές οικονομίες ε, ε, έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών επί τη βάση, ε, χωρών συγγνώμη, επί του επιμερισμού του, του βάρους, του άχθους. Ε, είναι σημαντικό να, δημιουργεί, να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία με την κατάλληλη μόχλευση θα μπορέσουν να μας δώσουν τα καλά αποτελέσματα. Να ε, ε, έχουμε πρόσβαση επίσης και στην ιδιωτική χρηματοδότηση. 40 εκατομμύρια ευρώ έχουν χρησιμοποιηθεί από ιδιωτική χρηματοδότηση στις 40 ενδιαφερόμενες χώρες και πολλαπλασιάστηκαν μέσω της μόχλευσης διαβούλευσης επί 40. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ε, καθολικό πλαίσιο ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε τους, τα, τείχη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Τρίτο και σημαντικό και τελευταίο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι να δημιουργηθούν εταιρικέ σχέσεις σωστές. Στο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μονάχα από την διακυβέρνηση θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο και η κοινωνία των πολιτών όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του θεματολογίου. Θέλουμε ε, να ε, υπάρξει ταυτόχρονα με το, ε, το πρόγραμμα τούτο και ένα, ένα, σημαντικό πλαίσιο λογοδοσίας που θα το στηρίζει. Η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα είναι επίσης ε, ιδιαίτερα ε, κρίσιμο, πολύ σημαντικό και ξέρω ότι και για το δικό σας κοινοβούλιο και για τα, και για τα ε, εθνικά κοινοβούλια αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερος προσφυλές. Ε, όσον αφορά δε την ε, έκθεση της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει, ε, να δώσει ένα πολύ καλό input όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και την γενικότερη συζήτηση επί του πλαισίου αυτού. Ευχαριστώ. Thank you very uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ε, σφαιρική προσέγγιση του θέματος και νομίζω ότι είστε έτοιμος να απαντήσετε και σε ερωτήσεις. Θα ήθελα βέβαια να σχολιάσουν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι μας το θέμα αυτό. Από το Eurodesk λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Jess Critchett σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να λάβω το λόγο εδώ. Θα αρχίσω με το γεγονός που συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Περέιρα και με τον Επίτροπο κύριο Μίμητσα η διάσκεψη είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο λόγω του θέματος που πραγματεύεται, αλλά και της χρονικής στιγμής ε, δηλαδή, είναι πριν από τη διάσκεψη του, 20, του 2015 και πριν από τη διάσκεψη στην αλλαγή του κλίματος και η επιτυχία των δύο επόμενων αυτών διασκέψεων του ΟΕΕ εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της διάσκεψης στην Αντισαμπέμπα. Αν εκεί πετύχουμε καλά αποτελέσματα και για το 2015 θα βοηθηθούμε και για την αλλαγή του κλίματος και αν αποτύχουμε στην Αντισαμπέμπα ε, αναλόγως θα αποτύχουν και οι επόμενες ε, διασκέψεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε καταρχήν ε, τι θα συμβεί στη Σύνοδο των λιγότερων επιτυγμένων χωρών πριν δούμε τι θα αποφασίσει η διευρυμένη G7 να μιλήσω για την ανακοίνωση που διάβασα για το συγκεκριμένο θέμα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να σας πω πως για την ανακοίνωση είναι μάλλον αντιφατικές οι απόψεις μου. Δηλαδή υπάρχουν δύο δυνατότητες να αναγνωριστεί ως είτε κάτι πολύ απογοητευτικό είτε ως μια πολύ επικίνδυνη στρατηγική. Απογοητευτικό γιατί είναι ελάχιστες οι συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει το θεματολόγιο αυτό. Εάν όντως αυτή είναι η αφιτηρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Ενδεχομένως όμως αυτό αποτελεί διαπραγματευτική τακτική. Δηλαδή καλύπτουν τις πραγματικές τους επιδιώξεις. Οπότε πιστεύω ότι η στρατηγική που ακολουθεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ούτε έξι μήνες δεν έχουν μείνει μέχρι την Αντισαμπέμπα χάνουμε πολύτιμο χρόνο σε μια στιγμή που θα έπρεπε εμείς να συνεργαζόμαστε με τα αναπτυσσόμενα κράτη για τα θέματα τα οποία τα ίδια θα ήθελαν να προσθέσουν στο θεματολόγιο της Αντισαμπέμπα. Έχω τέσσερα ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι θα είναι κρίσιμη σημασίας και για την διακυβέρνηση, την ομάδα G77 στον ΟΗΕ και για τις 150 οργανώσεις των της κοινωνίας των πολιτών παρουσιάσαν ένα έγγραφο στα τέλη της περσινής χρονιάς που ζήτησαν να είναι φιλόδοξα τα αποτελέσματα στην Αντισαμπέβα. Φορολογία. Ιδιωτική χρηματοδότηση. Βοήθεια και χρέος. Είναι λοιπόν αυτά τα κρίσιμα καυτά σημεία που εντοπίζω. Για τη φορολογία, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε από την αντισαβέβα είναι μια κυβερνητική φορολογική επιτροπή. Σίγουρα όλοι αναγνωρίζετε τη σημασία αυτού του θέματος. Και ξέρετε πως εμείς στη Eurodat κάναμε μια έρευνα πέρσι και προσπάθαμε να συγκεράσουμε όλες τις εισρωές κεφαλαίων προς τα ε, αναπτυσσόμενα κράτη και ε, να δούμε πόσα είναι όλα αυτά και είπαμε για κάθε ένα δολάρι, δολάριο ε, βοήθειας που μπαίνει στα ε, κράτη αυτά 97 cents ξαναφεύγουν παρανόμως. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα και φοροδιαφυγής αλλά και φοροαποφυγής. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε τα δύο θέματα αυτά μαζί στην αντισαβέβα, τότε δεν θα σημειώσουμε πρόοδο. Αυτή τη στιγμή η... ο τόπος στον οποίο συζητώνται τα θέματα αυτά είναι ο ΩΣΑ. Λάθος κατά τη γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό αποκλεί την πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων χωρών. Και αν σκεφτεί κανεί πω στον πυρήνα το προβλήματο τη ε, φοροδιαφυγή και τη φοροπολογή είναι η φορολογική παράδειση, τι μήνυμα στέλνουμε στι χώρε αυτέ, εάν δεν μπορούν καν να μπουν στη συζήτηση. Τι ενθαρρύνουμε. Τι ενθαρρύνουμε να θεωρούν πω είναι εκτό συστήματο, το οποίο ακριβώ είναι ο τόπο στον οποίο κρύβονται η φορολογική παράδοση. Δηλαδή, ε, ενθαρρύνοντά του να μην μπουν στην παγκόσμια συζήτηση για το θέμα αυτό, τη σωθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχουν και φορολογική παράδειση, για παράδειγμα ε, κάποιες, ε, κάποια βρετανικά εδάφη, το Λουξεμβούργο, ε, η Ελβετία, το Νόσα Αλλά παρόλα αυτά στις φορολογικές διαπραγματεύσεις χρειαζόμαστε μια διακυβερνητική επιτροπή σε επίπεδο ΟΗΕ. Η πρόταση αυτή στηρίζεται και από την G77. Είναι στο έγγραφο το οποίο παρουσίασε σχετικά ο ΕΕ για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και στηρίζεται από μια πολύ μεγάλη συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και φαντάζομαι θα μπορούσε να το στηρίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η δική σας κοινοβουλευτική έκθεση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, φορολογία. Το δεύτερο που είναι η ιδιωτική χρηματοδότηση, εδώ νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε τους όρους της συζήτησης. Η ιδιωτική χρηματοδότηση εισραίει στις αναπτυσσόμενες χώρες με υψηλούς κινδύνους, αλλά και πολύ υψηλά ε, ενδυνάμει αποτελέσματα. Και κίνδυνοι αυτοί πολύ συχνά αφήνονται στην άκρη, παρόλο που η G77 αναφέρεται στο γεγονός πως οι κίνδυνοι αποτελούν ακριβώς τον πυρήνα αυτών που τους ανησυχούν. Γι' αυτό και η ικανότητά τους να διαχειριστούν αυτή την ιδιωτική χρηματοδότηση πραγματικά ε, τις απασχολεί. Από το 2009 και μετά, σαν παράδειγμα να σας πω, πιο πολλά χρήματα έφυγαν από τις ε, χώρες αυτές ε, ως επαναπατρισμό κεφαλαίων ξένων επενδυτήσεων παρά ε, κεφάλαια από χρήματα που εισέρευσαν από ξένες επενδύσεις στις χώρες αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως επειδή ακριβώς υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών και, και όπω επίση και χρηματοστηρίων, καταλαβαίνετε πω η διαχείριση του κινδύνου που γίνεται από αυτά τα κράτη είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και πρέπει να μπει στο κέντρο των συζητήσεων. Όμω, όταν ξεκινάμε τι συζητήσει για την ιδιωτική εξωτερική χρηματοδότηση, σε τέτοιου είδου βήματα πολύ συχνά τελικά μιλάμε μόνο για το πώς μπορούμε να ε, προσελκύσουμε περισσότεροι ε, περισσότερες ξένες επενδύσεις στις χώρες αυτές. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της συζήτησης. Και αν δεν μιλήσει κανείς για το κίνδυνο, τα χρήματα αυτά να ε, φύγουν εκτός χώρας αμέσως, τότε αφήνει στην άκρη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του θέματος. Άρα λοιπόν, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό, ένα μείγμα βοήθειας για μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, τότε καταρχήν θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιδόσεις μέχρι σήμερα. Νομίζω πως ε, συνήθως έχουμε ιδιαίτερα διαφανή χρηματοδότηση που δεν έχει μεγάλη επιπτώσει στην ανάπτυξη και πηγαίνει κυρίως σε χώρους που είναι μέσω εισοδήματος. Δηλαδή δεν έχει δοκιμαστεί αυτό. Και επειδή υπάρχει μια τεράστια απώλεια, αν ε, χρησιμοποιήσει κανείς αναπτυξιακά κονδύλια για να κάνει κάτι τέτοιο, τότε χάνει αναπτυξιακά κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Εάν διαβάσετε και αν κοιτάξετε τι οδηγεί τι επενδύσει στα, στα αναπτυσσόμενες χώρες, θα δείτε πως θέλουμε να είναι υγιεί, ε, υψηλά εκπαιδευμένα ε, εργατικά σώματα, ε, χώρες, εγχώριε αγορέ αγορές κτλ. Και αυτό βεβαίω εξαρτάται και από τι δημόσιες υπηρεσίε που προσφέρουν οι δημόσιε επενδύσεις. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ μια παραδοσιακή στοχεύση που θα ήταν πιο χρήσιμη, δηλαδή επένδυση σε δημόσιες υπηρεσίες και δομές. Για το χρέος έχουμε εδώ μια μοναδική ευκαιρία φέτος να προχωρήσουμε. Να έχουμε μια μόνιμη πρόοδο στη λύση του προβλήματος του χρέους. Ξέρετε πως το 2012 οι ανεψόμενες χώρες έφτασαν στο υψηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο χρέους που είχαν ποτέ. Η Παγκόσμια Τράπεζα λέει 4,83 και έχουμε χώρες ε, που είναι χαμηλού εισοδήματο, που έχουν τεράστια προβλήματα ή είναι πολύ κοντά στην επικίνδυνη ζώνη με το χρέο του. Ευτυχώ κάποιε λύσει είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στον ΟΗΕ με μια διαδικασία για ένα πολυμερέ πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του εθνικού χρέου και ε, θα κλείσουν εκεί οι εργασίε μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντο έτου, αλλά δυστυχώ οι ευρωπαϊκέ χώρε αντέδρασαν πολύ καθυστερημένα στο θέμα αυτό και είτε απέχουν από την όλη διαδικασία, είτε δεν παίρνουν θέση. Και ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώ μπορεί αυτή η κρίση χρέου να διαιωνίζεται και να δημιουργήσει και να ζημιώσει πολύ τι οικονομίε. Εσεί λοιπόν θα μπορούσατε να παίξετε κάποιο πολύ θετικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Και τέταρτον, για την βοήθεια την ίδια, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Η βοήθεια είναι ακόμα πολύ σημαντική. Για χώρε χαμηλού εισοδήματο η βοήθεια είναι γύρω στο 10% ακόμα του ΑΕΠ. Είναι λοιπόν ένα κρίσιμο σημείο, ένα κρίσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Βέβαια, το 0,7 που είναι ο στόχο δεν πρόκειται να συζητηθεί. Θα επιβεβαιωθεί στην Αντισαμπέμπα και όλοι το γνωρίζουν. Όλε οι διαδικασίε του ΟΗΕ επιβεβαιώνουν αυτό το ποσοστό. Το ζήτημα είναι Υπάρχουν καλύτεροι μηχανισμοί για να εξασφαλίσουμε πως οι στόχοι αυτοί ε, ε πληρούνται. Δηλαδή, από το 2005 και μετά είπαν τα ευρωπαϊκά κράτη 0,7. Είμαστε στο 2015 και όπως είπε και ο Επίτροπος, ούτε στα μισά του δρόμου δεν έχουμε φτάσει. Έχουμε λοιπόν δεσμευτικού στόχου. Μπορούμε να του τοποθετήσουμε και στην ποιότητα τη βοήθεια. Δηλαδή να έχουμε μία απόζευξη όλη τη βοήθεια, γιατί βέβαια η βοήθεια αυτή όταν ε, είναι. Ε, όταν είναι συνδεδεμένη, μειώνει την απόδοσή της κατά 25%. Αποσύνδεση λοιπόν της βοήθειας, αποσυνδεδεμένη βοήθεια είναι αυτό που προτείνω. Αυτά από μένα και ελπίζω κάποια από αυτά να τα ακούσετε με θετικό πνεύμα και πιστεύω πως πραγματικά έφτασε η στιγμή να αυξήσει η ταχύτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες προτάσεις και να προχωρήσει στην κατεύθυνση της δέσμευσης και κυρίως μια διακυβερνητική επιτροπή για τη φορολογία, μια αλλαγή για τη συζήτηση που κάνουμε και τον τρόπο που συζητάμε τη ιδιωτική χρηματοδότηση για να δούμε ότι έχει και κινδύνους εκτός από ε, θετικά αποτελέσματα, ένας μηχανισμός για το χρέος για να κλείσουμε τα θέματα αυτά και κάποιους δεσμευτικούς στόχους για το ύψος βοήθειας. Thank indeed. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Θα συζητήσουμε τις προτάσεις σας σε λίγο. Θα ήθελα να περάσω τώρα στον κύριο Chris West. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πιστεύω πως όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, μάλλον έχω έρθει εδώ για να σας δώσω την, ε, την οπτική γωνία των ε, ιδιωτών του ιδιωτικού κεφαλαίου στο θέμα της αναπτυξιακής χρηματοδότησης και θα προσπαθήσω λοιπόν να πλησιώσω τις σκέψεις μου ε, αναφέροντας τους κινδύνους των ιδιωτικών επενδύσεων στην αναπτυξιακή βοήθεια αλλά αναφέροντας και τις ευκαιρίες που ενδεχομένως υπάρχουν και υπάρχουν όντως στον χώρο και ελπίζω να πυροδοτήσω ανταλλαγή απόψεων και συζητήσει από εσά. Τώρα, Είπα πως ήθελα να πλαισιώσω τα ε, σχόλιά μου. Θα ήθελα να σας πω ότι ανήκω στο Ίδρυμα Shell, που είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση η οποία διαχειρίζεται ιδιωτικό κεφάλαιο και λειτουργεί κάπως διαφορετικά από τις παραδοσιακές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Προσπαθούμε να δώσουμε λοιπόν απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις που έχουμε σχετικά με την ανάπτυξη ε, πρόσβαση σε νέες θέσεις απασχόλησης, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενεργειακά ζητήματα και είμαστε μία ένα ίδρυμα που έχει επιχειρηματική προσέγγιση. Και τι εννοώ με αυτό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα με εταίρους οι οποίοι δέχονται να μοιραστούν μαζί μας το ε, κίνδυνο καθώς και τους ε, στόχους αυτών των λύσεων που θέλουμε να δώσουμε, των βιώσιμων λύσεων δηλαδή. Εμείς παρέχουμε ένα μείγμα Επιχειρηματική στήριξης, χρηματοδότησης, εγγύηση ιδιωτικών επενδύσεων, συνδέσεων και συνεργασιών με άλλους εταίρους και φυσικά συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας και παρακολουθώντας τις επιδόσεις, θέτουμε στόχους επιδόσεων και βοηθούμε τους εταίρους μας στις προσπάθειές τους να συγκεντρώσουν μοχλευμένο κεφάλαιο, όχι μόνο ιδιωτικό αλλά και δημόσιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να γίνουν ανεξάρτητοι. Αυτή η προσέγγιση νομίζω πως μας οδήγησε στην επιλογή λίγων οργανώσεων οι οποίες ασχολούνται ακριβώς με αυτές τις αναπτυξιακές προκλήσεις στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και προσπαθούν να έχουν ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ίσως ε, να έχετε ακούσει τους όρους Venture Philanthropy και Impact Investing, επιχειρηματική φιλανθρωπία και επενδύσεις αντικτύπου δηλαδή. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια με τις ε, δράσεις μας έχουμε δημιουργήσει συνεργασίες με διάφορους φορείς, με κρατικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών, την επενδυτική του τράπεζα, οι οποίοι στηρίζονται σε μας για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν αυτούς τους ε, στόχους και αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Τώρα, όσον αφορά τους κινδύνους, να σας πω ότι σε νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα είναι δύσκολο να ε, υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Δεν υπάρχει η κατάλληλη ευελιξία και η κατάλληλη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση. Έπειτα, η πρωτη δικαιούχοι αυτών των νέων επιχειρηματικών μοντέλων δεν είναι οι φτωχότεροι. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει άμεσο αντίκτυπος στη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω αυτά τα νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα σπάνια δημιουργούν άμεσα ε, προοπτικές κέρδους. Γι' αυτό λοιπόν δύσκολα προσελκύουν άμεσα επενδυτές. Και εδώ έρχομαι να πω τις δικές μου προτάσεις για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα με τον ιδιωτικό τομέα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι όλο ένα και περισσότερο φιλανθρωπικό εντό κεφάλαιο απελευθερώνεται. Και παίρνει αυτό διάφορες μορφές και αφορά διάφορε ομάδε ανθρώπων. Και εδώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Μπορεί να κινητοποιήσει αυτό το φιλανθρωπικό κεφάλαιο έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα να επενδύσουν πάνω σε αυτές τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και παρέχοντάς τους βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Υπάρχουν ευρωπαϊκές ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό και προωθούν το φιλανθρωπικό κεφάλαιο για επενδύσεις. Και αυτό που χρειάζεται είναι να πιστούν αυτοί οι οργανισμοί να υιοθετήσουν καινοτόμε προσεγγίσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα παρά τις παραδοσιακές που είναι και πιο μακροπρόθεσμες. Πιστεύω πως έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία εδώ να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους για την ε, αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Έπειτα, αναφέρθηκα στους κινδύνους. Πιστεύω πως με την πάραδο του χρόνου ε, υπήρξε μια αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών ζητημάτων από την ε, παραδοσιακή, θα έλεγα, εταιρική κοινωνική ευθύνη προς την διοχέτευση πόρων για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συγκεκριμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα. Από την εταιρική κοινωνική ευθύνη δηλαδή πήγαμε στην κοινωνική εταιρική ε, ευκαιρία. Αυτό είναι κάτι θετικό για τον ιδιωτικό τομέα, παρότι είναι ρηψοκίνδυνο. Διότι ο ιδιωτικός τομέας επενδύει στην ουσία σε κάτι που δεν είναι τόσο σίγουρο όσο το παραδοσιακό μοντέλο. Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη σύνδεση και τη συνδεσιμότητα των διάφορων ε, χώρων. Για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα να καταλάβουν επισητιστικά ζητήματα και ζητήματα υγιεινής. Εάν δεν υπάρχει κάποια σαφή σύνδεση των στόχων, είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσεις ιδιωτικό κεφάλαιο. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι η αριστεία στον ιδιωτικό τομέα, στις ιδιωτικές επενδύσεις, χαρακτηρίζεται κυρίως από την καινοτομία. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε τις τραπεζικές συναλλαγές από κινητά τηλέφωνα. Αυτή είναι μια καινούρια τεχνολογία, όμως αυτή η τεχνολογία δεν θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί ε, μόνο από ιδιωτικά, ιδιωτική πρωτοβουλία. Χρειάζεται και η συνεργασία και η σύμπραξη του δημόσιου τομέα. Χρειάζεται λοιπόν καινοτομία, χρειάζεται, χρειάζονται νέες ιδέες και εμείς ως Ίδρυμα Shell έχουμε αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες και τώρα είμαστε πρωτοπόροι στην παροχή ενέργειας στις πιο φτωχές χώρες. Προσελκύουμε ιδιωτικό κεφάλαιο και το χρησιμοποιούμε για να αναπτύσσουμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο και μετά να επεκταθούμε και σε άλλες αγορές. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι επενδύσεις έχουν ένα ξεκάθαρο κοινωνικό όφελος, όμως δεν είναι άμεσα βιώσιμες. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η ευκαιρία για τον δημόσιο τομέα να βγάλει τον κίνδυνο από τους ε, ιδιώτες επενδυτές. Επίσης, τα καλύτερα επιχειρηματικά μοντέλα δείχνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στην δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Όμως η δική μου εμπειρία λέει ότι δεν ε, καταφέρνουν να δημιουργήσουν αρκετό κέρδος έτσι ώστε να γίνουν εμπορικά ελκυστικές. Και βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για μια ανάμεικτη χρηματοδότηση που είναι πραγματικά ζήτημα ζωής και θανάτου για μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε να κλιμακώσουμε τόσο μια ιδέα, μια επιχείρηση έτσι ώστε να προσελκύσει ιδιωτικό κεφάλαιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν το δημόσιο τομέα εδώ για να παρέχει αυτή τη δυνατότητα της ε, ανάμιξης του blending στη χρηματοδότηση. Να υπάρχουν δηλαδή κάποια δάνεια ε, τα μακροπρόθεσμα μετοχικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμα δάνεια και ε, καινοτόμες χρηματοδοτικές ε, δομές οι οποίες θα επιτρέψουν αυτά τα, αυτές τις νέες επιχειρήσεις, τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να τοπίσουμε αυτές τις κεφαλαϊκές δομές Προσπαθούμε, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε ένα ταμείο το οποίο θα στηρίζει τις νέες επιχειρήσεις, της startups στην Αφρική. Και έχουμε δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο ιδιωτικό κεφάλαιο με συνδρομή και κυβερνήσεων τη γερμανική κυβέρνηση για παράδειγμα, το οποίο διατίθεται ακριβώς σε αυτέ τι επιχειρήσεις οι οποίες από μόνες τους δεν είναι ε, δυνατόν να προσελκύσουν αμέσως ιδιωτικό κεφάλαιο. Πιστεύω λοιπόν πως υπάρχει τεράστιο δυναμικό και γι' αυτό χρειαζόμαστε δημιουργικά μυαλά. Τέλος, ε, θα σας αναφέρω την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πιστεύω πως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το κλειδί για την επιτυχία της σύμπραξης αυτής είναι ε, ο ξεκάθαρος στόχος της συνεργασίας αυτής. Χρειάζονται κοινοί λοιπόν στόχοι, ξεκάθαροι δείκτες επιδόσεων, ίσως καταμερισμός του κινδύνου σε όλους τους εταίρους, επαρκής χρηματοδότηση και ξεκάθαρες δομές για τη λογοδοσία και για τον έλεγχο των επιδόσεων. Έχουμε κάποια εξαιρετικά παραδείγματα, όπως για παράδειγμα στην έκθεση ΣΑΞ, και η δική μου εμπειρία δείχνει ότι τα προγράμματα αυτά αποτυγχάνουν όταν υπάρχει ε, αδυναμία λήψης αποφάσεων, όταν δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αφείς δομές και αδύναμα μοντέλα σύμπραξης δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Συμπερασματικά θα μπορούσα να πω ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει να προσφέρει πάρα πολλά στους ε, στόχους εφορίας για την ανάπτυξη και πρέπει να πάρουμε λοιπόν αυτή την επιχειρηματικότητα που έχει ο ιδιωτικός τομέας και να ε, βάλουμε την ασφάλεια του δημόσιου τομέα έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι το καλύτερο. Θα ήθελα λοιπόν λέγοντας αυτά να κλείσω λέγοντας ακόμα μια φορά ότι θεωρώ ότι η ανάμειξη αυτού του κεφαλαίου είναι εξαιρετικά σημαντική, αναγκαία για την επιτυχία του μοντέλου αυτού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είδαμε το ίδιο θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Είναι η ώρα των ερωτήσεων ε, και των απαντήσεων. Θα έχουμε λοιπόν μια μικρή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε όλους τους πανελίστες που πήραν το λόγο. Μία ερώτηση για τον Επίτροπο Μίμητσα. Ακούγεται και συζητιέται ότι το ODA είναι ένα μικρό τμήμα της ε, ανάπτυξης και της αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, μπορεί να υπάρξει, να είναι του, της τάξης του 1% ή μια, να υπάρξει και διπλασιασμός. Ξέρουμε ότι είναι ένα μικρό κομμάτι όμως της βοήθειας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έτσι ώστε ε, να μην ξεχωρίσουμε το ODA από άλλες ε, συζητήσεις δηλαδή να συνεχίσει και η συζήτηση για τους γενείς πόρους και για την, τους πόρους από κτλ γιατί διαφορετικά στην Αντίσαβέμπα ενδεχομένως δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ε, ε, καλή συζήτηση και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο και στις ε, συζητήσεις της Νέας Υόρκης αλλά και του Σεπτεμβρίου μετά αλλά και του Δεκεμβρίου στο Παρίσι για το κλίμα. Απ' την άλλη πλευρά δημιουργήσουμε ε, μια, ένα καλό περιβάλλον ας πούμε ε, όπου θα δείχνουμε την καλή μας θέληση στην Αντίσα Μπέμπα ενδεχομένως ε, αυτό θα έχει καλό αντίκτυπο και σε όλα τα υπόλοιπα γιατί υπάρχει διασύνδεση μεταξύ όλων των συναντήσεων. Εμείς έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά με τους συναδέλφους μας των χωρών ΑΚΕ αλλά οπωσδήποτε στην Αντίσα Μπέμπα πρέπει να βγάλουμε όλα τα χαρτιά μας και να τα βάλουμε στο τραπέζι. Πώς βλέπετε να προχωράει το θέμα όσον αφορά το 0,7% λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ευρώπης. Ε, θα είναι δύσκολο το 0,7%. Τζες, αναφέρθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, ο Κρίς μάλλον το είπε αυτό. Ε, μας έδωσε την άποψή του για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό, ιδιωτικό τομέα. Πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος ε, πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει απλώς το προπέτασμα καπνού έτσι ώστε να, να, ε, κάνουν επενδύσεις ας πούμε οι ε, ιδιωτικές εταιρείες με δημόσιο χρήμα. Θέλω παράδειγμα, πες μου, αυτό έγινε εκεί και αυτό. Ε, λειτουργήσε, δεν λειτουργήσε. Ίσως είναι λίγο προκλητικό αυτό που θα πω τώρα. Μίλησες για τον ιδιωτικό τομέα ε, και τον δημόσιο τομέα ε, που θα πρέπει να μοιραστεί τον κίνδυνο, να μοιραστούν τον κίνδυνο. Ε, εγώ θα το αντέστρεφα. Θα έλεγα μήπως ο ιδιωτικός τομέας θα μοιραστεί τα κέρδη. Στην Ευρώπη γίνεται μεγάλη συζήτηση, γίνεται μεγάλη συζήτηση και για το ευρώ κιόλα ε, ε, και για τα, για τα χρήματα που, για το ευρώ το οποίο δεν βοηθάει τις ιδιωτικές επενδύσεις κτλ. Ε, στις χώρες που δουλεύεις βλέπεις επιστροφή μέσω φόρων και αν ναι σε τι επίπεδο. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρούιμπιχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτή η ακρόαση έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι δηλαδή μπορούμε από τώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον. Και πιστεύω ότι μια που βρισκόμαστε στο έτος ανάπτυξης, Πρέπει να δημιουργήσουμε και τις αναγκαίες δομές για αυτή. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος ΣΕΛ σχετικά με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Ποιο ρόλο παίζουν οι παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις και πώς μπορούμε αυτές τις ε, οικογενειακές επιχειρήσεις να τις ε, οθήσουμε να δημιουργήσουν δομές ή να ενταχθούν σε υφιστάμενες δομές έτσι ώστε να ε, αναπτυχθούν. Και τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές δομές. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Πέντρο. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο για να πούν τόσο ενδιαφέροντα πράγματα πλήρη εναυσμάτων. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι η συζήτηση αυτή θα μας οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στην αντίσαμπέμπα και θα την συνεχίσουμε βεβαίως όχι μόνο σε σχέση με την έκθεση για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αλλά ε, και μέσω μιας έκθεσης ε, ε, για το θέμα το οποίο έθιξε ο εκπρόσωπος της Eurodebt όσον αφορά την φοροδιαφυγή και τα έσοδα τα φορολογικά, γιατί υπάρχει μεγάλη διασύνδεση. Ε, ο Επίτροπος αναφέρθηκε σε φορολογικά συστήματα που πρέπει να είναι πιο σαφή, πιο δίκαια και βεβαίως ε, και ε, πρέπει εδώ να γίνει αναφορά και στις παράνομες, στην ροή παράνομου χρήματος τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι συγκλονιστικά ε, και δείχνουν πόσο αυτού του είδους ε, τα προβλήματα μπορούν να δυναμητήσουν και την προσπάθειά μας ε, και την ανάπτυξη γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν νέα εργαλεία και νέες λύσεις έτσι ώστε Ε, τα θέματα της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής ε, να μπορέσουμε να ε, κάνουμε σημαντικά βήματα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα σεμινάριο. Πολλοί μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας εδώ θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό που θα έχει ακριβώς τα, θέματα τα φορολογικά στο επίκεντρό του. Έχουμε μπροστά μας πολλές ημερομηνίες σημαντικές. Έχουμε την Αντίσα Μπέμπα, έχουμε ε, αυτό το νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη μετά το 2015. Έχουμε τη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Εάν η Αντίσα Μπέμπα δεν μπορέσει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα, τότε ενδεχομένως θα αποδυναμωθούν ε, και τα, ε, ε, οι κατοπινές συνεδριάσεις στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι μπορεί να σπρώξει προς την κατεύθυνση μιας πιο φιλόδοξης ε, λύσης. Αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει η ανάμειξη να είναι μεγαλύτερη, θα πρέπει να ξεπεραστούν ε, κάποιες ακαμψίες και ελπίζω να το κάνει αυτό η Επιτροπή γιατί θα βοηθήσει και τον εαυτό της και εμάς όλους στη δικιά μας δουλειά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάποιος από το κοινό θέλει να πάρει το λόγο, θέλει να ρωτήσει κάτι ε, τους ομιλητές μας, να αντιδράσει σε κάτι που άκουσε. Όχι. <coughs> από ό,τι βλέπω κανείς. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να υποβάλω δύο ερωτήματα. σε σχέση με αυτό το στόχο του 0,7%. Το θέμα είναι τεχνικό ή είναι κάτι περισσότερο. Καταλαβαίνουμε ότι η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση η οποία στόχο, η οποία ε, θα έπρεπε ε, τελικά να εγκριθεί από το Συμβούλιο, από τα κράτη-μέλη δηλαδή. Καταλαβαίνουμε όλοι τη δυσκολία του εγχειρήματο. Όμως, το ερώτημα είναι το εξή. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, για να έχουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι η οδός που προτείνει η Κομισιόν στόχος 0,7, στήριξη και η συζήτηση να γίνει με όλους τους εταίρους για μια γενική συμφωνία ή θα πρέπει να είναι εμβληματική ας πούμε η πρόταση παραδειγματική ε, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ίδιο ε, ε, μηχανισμό επιθεώρησης και παρακολούθησης κτλ. Αυτό είναι στρατηγική σημασία θέμα και ε, οπωσδήποτε αφορά άμεσα την διάσκεψη της Αντισαμπέμπα. Γιατί αν θέλουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο, ηγετικό ρόλο στην Αντίσα Μπέμπα, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες στρατηγικές επιλογές. Θα ήθελα ο Επίτροπος να μου απαντήσει πάνω σε αυτό. Δεύτερον, η διάσκεψη της Αντίς Αμπέμπα είναι, σε επίπεδο, είναι πρεσβευτικού επίπεδου, όπου θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Επομένως θα υπάρχουν και λόγοι, θα υπάρχουν ε, προφορικοί, θα υπάρχουν όμως και γραπτά έγγραφα. Στο τέλος περιμένουμε να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις. Ας πούμε, λέμε ότι τα μηνύματα είναι σημαντικά, λέμε ότι η βελτίωση ας πούμε του φορολογικού συστήματος είναι θεμελιώδου σημασίας και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ε, διεθνή συνεργασία. Ερώτημα. Ποια θα είναι η πολιτική απόφαση η οποία θα ληφθεί στην Αντίσα Μπέμπα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Πολιτική απόφαση, για πολιτική απόφαση μιλάμε. Γιατί τώρα μία γενικόλογη δήλωση βάσει της οποίας ε, έχουν μεγάλη σημασία τα φορολογικά συστήματα είναι ωραία, σημαντικό, αλλά δεν περιλαμβάνει πολιτική δέσμευση. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πώς ε, βλέπει τα πράγματα. Υπάρχει δυνατότητα, είναι πιθανό να υπάρξει πολιτική απόφαση, υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές που ανοίγονται μπροστά μας. γιατί καλά τα λόγια, αλλά θέλουμε και έργα. Όσον αφορά δε την συνολική διακυβέρνηση, global governance. Τι περιμένετε να γίνει στην Αντίσα Μπέμπα. Ωραία, θα δώσω τώρα ξανά το λόγο στους ομιλητές, στο πάνελ. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Εσείς αποφασίστε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές ερωτήσεις. Ε, αυτές κυρίως ε, για το φορολογικό σύστημα και τη γενική χρηματοδότηση. Έχετε δίκιο που το ρωτάτε τι είδους απόφαση μπορεί να ληφθεί ή τι είδους αποφάσεις μπορούν να ληφθούν στην Αντίσα Δεν μιλάμε για διακυβερνητική ε, διάσκεψη, επομένως ε, αποφάσεις οι οποίες προωθούν ε, τα θέματα πραγματικά είναι, ε, και δίνουν συνέχεια είναι πολύ σημαντικές γιατί με τον τρόπο αυτό ξεκινούν σημαντικές συζητήσεις ας πούμε για να γίνει το Διεθνές Φορολογικό Σύστημα πιο δίκαιο για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Επίσης μπορούν να υπάρξουν δεσμεύσεις επί άλλων ε, ε, στόχων και επί της καλύψεως άλλων στόχων με δεσμευτικό τρόπο. Πολλά μπορεί να πετύχει κανείς. Βεβαίως και γι' αυτό ακριβώς εμείς θέλουμε να δούμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να παίρνουν μία ε, πιο ενεργητική στάση και να παίζουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο ε, ε, ε, γενόμενοι ηγέτιδες ας πούμε δυνάμεις και δείχνοντας το δρόμο δια του παραδείγματος. Να δούμε τι κάνουν οι τράπεζες με τα χρήματά τους, πώς τα χρησιμοποιούν, πώς τα επενδύουν κτλ. Νομίζω ότι αυτό τώρα έφτασε η στιγμή για να ε, ανοίξουν και τα κεφάλαια αυτά και να γίνει αυτή η συζήτηση που θα είναι ε, σημαντική και για όλα τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να αλλάξουμε το κλίμα στην Αντίσα Μπέμπα. Νομίζω ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε. Όσον αφορά τώρα την ιδιωτική χρηματοδότηση. Μπορώ να συμφωνήσω με τον κρίση, ίσως για όχι για τους ίδιους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους μακροοικονομικούς κινδύνους και τους μικροοικονομικούς. Η μακροοικονομική είναι πολύ σημαντική διάσταση για τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες ε, εδώ και 100 χρόνια οι χώρες αυτές ε, αντιμετωπίζουν ε, ε, κρίση δημοσίου χρέους και ε, πολύ συχνά οι χρηματοδοτικές κρίσεις ε, που είναι απόρρια των, ε, του δημόσιου χρέους και της κατάστασης του δημόσιου χρέους μπορούν να πυροδοτήσουν μεγάλες και σοβαρές κρίσεις σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως, εάν δεν καταφέρουν οι χώρες να ελέγξουν καλά την εισρωή, εκροή κεφαλαίων κλπ, τότε ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν είναι ε, πολύ ε, μεγάλος. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι όμως και ξέρουμε πολλά ε, παραδείγματα ε, ξένων επενδυτών που μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν την δύναμή τους καθώς επίσης και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών έτσι ώστε να πετύχουν ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, φορολογικές εκπτώσεις, διαφορετικό ας πούμε κοινωνικό περιβάλλον και οικονομικό ε, αντίκτυπο κτλ. Έχουμε πολλά παραδείγματα ε, για επενδύσεις οι οποίες ε, έχουν εν τέλει τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παρόλα αυτά έχουν βρει συμφωνίες με τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών. Ε, απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα το ερώτημα που τίθεται είναι πώς ε, θα υπάρξει κινητροδότηση έτσι ώστε κάποιες εταιρείες να ενδιαφερθούν να ε, πάνε στις περιοχές αυτές. Υπάρχει το ζήτημα της μεταφοράς του κινδύνου που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα ε, Ένας τρόπος αντιμετώπισης θα ήταν ας πούμε αυτός που αναφέρατε προηγουμένως, ε, δηλαδή ε, οι δημόσιες επιδοτήσεις, επιδοτήσεις μέσω του δημοσίου. Επίσης υπάρχουν τράπεζες όπως η Τράπεζα Γεωργικής Ανάπτυξης που μπορούν να αναλάβουν τέτοιου είδους κινδύνους έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι απαραίτητες επενδύσεις θα γίνουν στον κατάλληλο, στην κατάλληλη περιοχή το 2012 ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες είχαμε 35%, 35 ε, του ΑΕΠ ε, αυτής οι επενδύσεις. Οι, οι μεδαπές επενδύσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όταν μιλάμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες το ερώτημα δεν τίθεται ε, επί τη βάση του ε, ποια κίνητρα μπορούν να δώσουν έτσι ώστε να γίνουν σωστές επενδύσεις. Ε, η συζήτηση συνήθως γίνεται για τα χρήματα, για, την, για τις επιδοτήσεις, για το δημόσιο χρήμα που μπορεί να επιτευχθεί κτλ. Επομένως, συμφωνώ, συμφωνώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενθαρρύνουμε τους ε, επενδυτές αλλά στα πλαίσια της ε, ιδιοκτησίας που θα παραμένει στα χέρια των τοπικών κυβερνήσεων, των, τοπικών, των χωρών. Ε, Κρίστελ, να πεις ε, και εσύ κάτι, ίσως να σχολιάσεις και το τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα με τους, ε, με τα, τους επενδυτικούς στόχους. Λοιπόν, θα απηχήσω τόσο, όσα είπε ο Τζέσι και για τους κινδύνους που ελοχεύει η χρηματοδότηση από ιδιωτικά κονδύλια. Ε, διαχειριζόμαστε λοιπόν ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό κάνω. Ε, τα οποία ε, εμφανίζονται ως φιλανθρωπικές ε, οργανώσεις. Άρα λοιπόν είναι φιλανθρωπικά κεφάλαια τα οποία εξεργαμίζονται πολύ με τις προσπάθειες που κάνουμε για τις δημόσιες επενδύσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε, πώς θα μεγιστοποιήσουμε ότι τα ιδιωτικά κέρδη θα είναι μία απλή επίπτωση ε, παράλληλα με, τις δημο... με, τα... με τα κέρδη για το δημόσιο, γιατί ως φιλανθρωπική οργάνωση είμαι υποχρεωμένος να μετρήσω ε, καταρχήν αν θα προκύψουν κάποια κέρδη και πόσο θα είναι αυτά. Η δική μου εμπειρία μου λέει πως όταν έχουμε χρηματοδοτήσει ε, κοινωνικές επιχειρήσεις ε, κερδοσκοπικές, οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι πολύ ευρύτερες από αυτές σε σχέση με τις αντίστοιχες φιλανθρωπικές οργανώσεων. Και πρέπει να πω ότι τα κέρδη στην περίπτωση αυτή είναι πολύ μικρά γιατί ε, δεν είναι αυτή η στόχευση των έργων που επιλέγονται. Άρα λοιπόν η εμπειρία μου στον κλάδο αυτό μου λέει πως μπορεί κανείς να διαχειριστεί και να μετρήσει ε, στο πακέτο βοήθειας ακριβώς πώς θα γίνει αυτή η κατανομή. Κάποιες από τις κοινωνικές επιχειρήσεις που τώρα αναδύονται είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος με τις καλύτερες θετικές επιπτώσεις για να φέρουν την κοινωνική αλλαγή και ε, ελαχιστοποιούν ε, την, ε, τον κίνδυνο των ιδιωτικών κερδών που θα εκπατριστούν η βασική φιλανθρωπία έχει διαφορετική στόχευση και ένα από τα προβλήματα τα οποία ιστορικά αντιμετωπίζει ο κλάδος φιλανθρωπίας είναι πως βασίζεται σε βράχη πρόθεσμη χρηματοδότηση η οποία περιορίζεται στην διάρκεια και περιορίζεται στη στήριξη μόνο συγκεκριμένων φιλανθρωπικών δράσεων το οποίο σημαίνει ότι η πλειοψηφία των φιλανθρωπικών οργανώσεων δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το ίδιο τους το κέρδο και χάνουν πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να βρουν ε, χρήματα για να καλύψουν τα λειτουργικού τα λειτουργικά τους κέρδη και δεν μπορούν να βρουν τα κεφάλαια που θα τους επιτρέψουν να μεγαλώσουν και να λειτουργήσουν σωστά με αποτέλεσμα να μην δίνουν πάντα τα θετικά αποτελέσματα που χρειάζονται. Και όταν μιλώ για επιχειρηματική φιλανθρωπία, μιλώ για προσπάθειες που γίνεται αυτές τις οργανώσεις να τις οικοδομήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο που θα μπορούν οι ίδιες να παρέχουν και τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα χωρίς να στοχεύουμε σε συγκεκριμένα έργα κάθε φορά αλλά πρικοδοτώντας με πόρους για να μπορούν να απελευθερωθούν από το συνεχή περιορισμό να ψάχνουν κεφάλαια και να έχουν την δυνατότητα να ε, εκτελέσουν το φιλανθρωπικό τους έργο με αποτελεσματικό τρόπο. Άρα λοιπόν μιλώ για φιλανθρωπική επιχειρηματικότητα ή για φιλανθρωπικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης δράσης και μετά να μπορούν να επιστρέψουν στους δωρητές και να πούν μπορείτε να μας χρηματοδοτήσετε παραπάνω γιατί θέλουμε να κάνουμε και κάτι επιπλέον. Έτσι λοιπόν οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν θα έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για μένα η παραδοσιακή φιλανθρωπία είναι ένας ο τρόπος με τον οποίο παραδοσιακά οι δωρητές ε, χρηματοδοτούσαν κάποια ε, βραχυπρόθεσμα έργα. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ανεπτυξιακά προβλήματα, τότε θα πρέπει ο τρόπος που οικοδομούνται αυτές οι οργανώσεις να είναι πιο επιχειρηματικός, έτσι ώστε να έχουν τις βασικές δυνατότητες και προσόντα να καλύψουν ακριβώς αυτά τα οποία χρειάζεται. Και τελικά, επειδή εγώ είμαι από μικρή επιχείρηση, πρέπει να πω πως πραγματικά κατανοώ ε, και επαναλαμβάνω τα όσα είπατε περί ε, σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα στις αναδυόμενες ή στις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλοί λένε πολυεθνικές αμέσως. Αλλά για μένα στις αναδυόμενες ε, χώρες το πιο βασικό είναι ο μικρομεσαίος κλάδος, ο οποίος ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου. Και η πρόκληση για τον κλάδο αυτό είναι να βρει κεφάλαια, κεφάλαια κίνησης. Η πραγματικότητα είναι όμως δεν είναι μόνο η έλλειψη επιχειρηματιών σε κανένα κράτος δεν λείπουν επιχειρηματίες. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζονται στήριξη, επιχειρηματικές ε, ε ικανότητες και γιατί δεν έχουν τις εγγύησεις που, ε, που χρειάζονται για να πάνε σε μια τράπεζα και να βρουν χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν χρειάζονται και ε, κεφάλαια ε, κινδύνου και μόνο μέσω αυτών θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την καινοτομία, την ανάπτυξη και είναι τόσο σημαντικό και για το δημόσιο κλάδο και για τον ιδιωτικό κόσμο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί στον ιδιωτικό κόσμο δημιουργεί θέσεις εργασίας, διαφοροποίηση ε, στον κόσμο των επιχειρήσεων και στο δημόσιο κλάδο για τους λόγους που μόλις παρουσίασα. Γι' αυτό είναι εύκολο λοιπόν να εντοπίσουμε τα προβλήματα, πρόσβαση σε ικανότητες, πρόσβαση σε κεφάλαιο, και το ζήτημα είναι να προσφέρουμε επιχειρηματικέ λύσει στι προκλήσει αυτέ που θα εντάξουν στο μοντέλο αυτό και σε αυτό το μερίδιο τη αγορά και τα επιχειρηματικά προσόντα και τα επιχειρηματικά κεφάλαια που χρειάζονται, έτσι ώστε να υπάρχει και κάποιο περιθώριο κέρδου για να μπορούν οι εταιρείε αυτέ μέσα στα επόμενα χρόνια να μεγαλώσουν κιόλα. Υπάρχουν οι φορεί τη ε, της που μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, επειδή ακριβώς το πρόβλημα του κέρδους υπάρχει, επαναλαμβάνομαι ότι γι' αυτό στήσαμε αυτή την εταιρεία στην Αφρική για να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, αλλά χρειαζόμαστε ένα διακεκομένο σύστημα που θα επιτρέψει να έχουμε αυτό το μείγμα το οποίο ε, θα είναι κυλιόμενο και θα μας επιτρέψει να τροφοδοτούμε όλη αυτή την προσπάθεια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα σημαντικός κλάδος και νομίζω το είπατε κι εσείς. Χρειάζεται να πάρουμε τον κόσμο από την άτυπη οικονομία που έχει να κάνει με την επιβίωση και να τους εντάξουμε στον, στην επίσημη οικονομία που πληρώνει φόρους, που καταγράφεται και μετά μπορούμε να δούμε πώς λογοδοτούμε για τα κέρδη τα οποία ε, δημιουργήθηκαν κτλ. Αλλά σίγουρα 100% ο κλάδος των μικρομεσαίων είναι ο τόπος συνάντησης του ιδιωτικού και του δημόσιου ε, και της δημόσιας χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει λοιπόν το πάνελ αυτό με την παρέμβαση που θα κάνει ο Επίτροπος Μίμητσα. Να ξεκινήσω μιλώντας για το ποια είναι η φύση ίδια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω να μην έχασε κανείς ούτε μία γραμμή από τη δήλωσή μας, τη δήλωσή μου και κυρίως αυτή που λέει πως θα πρέπει αυτή η ανακοίνωση να μεταφραστεί σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Δηλαδή, υπάρχουν δύο διαδρομές διαπραγμάτευσης ενώπιών μας. Μία διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, πριν το Συμβούλιο και η άλλη διαδρομή θα ακολουθήσει τις ε, διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη και στην Μπέμπα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία έτσι ώστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να είναι φιλόδοξα και συγκεκριμένα. Θα πρέπει να φροντίσουμε η ανακοίνωση να αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων για τη θέση μας τη διαπραγματευτική και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Ίσως λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις ανοιχτά. Ίσως δεν μπορούμε να μιλήσουμε όσο ανοιχτά θα ήθελαν κάποιοι στην ανακοινωσή μας, αλλά σίγουρα εμείς θα βασιστούμε στην ανακοίνωση αυτή και στα επόμενα στάδια θα χτίσουμε πάνω στα όσα παρουσιάσουμε. Αυτό για τις επόμενες διαπραγματεύσεις που θα γίνουν όχι μόνο στο Συμβούλιο αλλά και με τους υπόλοιπους εταίρους. Τώρα για την Αντίσα Μπέμπα να σας πω τα εξής. Λυπάμαι. Γιατί είναι αρκετά σαφές και ανησυχώ και εγώ για το γεγονός πως όντως υπάρχει κίνδυνος στην Αντισαμπέμπα να συζητήσουμε μόνο ε, τις δικούς μας στόχους για την αναπτυξιακή βοήθεια εκτός Ένωσης. Και νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο στόχος ούτε ο δικός μας ούτε ο στόχος των κρατών μελών. Θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε ή εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς στο να αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος. Η δική μας ε, σφαιρική προσέγγιση συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα από την κλασική αναπτυξιακή βοήθεια που στέλνουμε στο εξωτερικό, ε, όχι μόνο γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις ε, στο επίπεδο του 0,7% του ΑΕΠ, ούτε γιατί προσπαθούμε να αναφερθούμε σε άλλα είδη χρηματοδότηση, αλλά γιατί πιστεύουμε πως αυτή η σφαιρική προσέγγιση, η συνολική προσέγγιση είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε το αναπτυξιακό θεματολόγιο και τις αναπτυξιακές ανάγκες των ε, χωρών ε, εταίρων μας. Ο στόχος του 0,7% τουλάχιστον σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις δικές μας προτάσεις και συστάσεις στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο, είναι ξεκάθαρος. Ας επαναδεσμευθούμε συλλογικά υπέρ του 0,7%. και ας αφήσουμε ένα περιθώριο στις διαπραγματεύσεις στο χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε ο στόχος αυτός να ενταχθεί στο χρονοδιάγραμμα και οι υπόλοιπε αναπτυγμένες ή ε, υψηλού εισοδήματος χώρες και οι βασικοί δωρητές να ε, συμβαδίσουν ε, με το στόχο αυτό μαζί μας. Πήγαμε και κάπως πιο μακριά στην ανακοίνωση τη δική μας και δεν προτείναμε μόνο να επαναδεσμευτούμε στο 0,7% αλλά είπαμε πως θα δεσμευτούμε υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας για τις λιγότερο για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που θα φτάνει υψηλότερα και από αυτό. Recalling the, the fact that nowadays there is Σήμερα είναι χαμηλότερο το επίπεδο των δεσμεύσεων και αυτό συμβαίνει ε, λόγω και της εισόδου νέων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε στο 0,33 νομίζω. Οπότε λέμε 0,7% συλλογικά θέλουμε να πετύχουμε. Για εμένα προσωπικά το θέμα αυτό δεν είναι απλά τεχνικό. δεν είναι θέμα μόνο δημοσιονομικής διαπραγμάτευσης. Δεν είναι θέμα απλά διαπραγμάτευσης συνεισφοράς των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον προϋπολογισμό αυτής. Όχι. Έχει να κάνει με την πολιτική δέσμευση που αναλαμβάνουμε. Είναι μια πολιτική κατεύθυνση που επιλέγουμε. Είναι ένας πολιτικός δρόμος που θα μας φέρει κοντύτερα στους στόχους μας την αναπτυξιακή βοήθεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ηγηθούμε εμείς μέσω του παραδείγματος που θα δώσουμε. Και πιστεύω πως όλοι χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι την συνειδρίαση του Συμβουλίου και τις διαπραγματεύσεις που θα κάνει για τον προϋπολογισμό, αλλά νομίζω πως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζομαι στο να σας περιγράψω τη δική μου άποψη και τη δική μου προσέγγιση. Αυτή η στάση που προτείνω, δηλαδή να ηγηθούμε μέσω του παραδείγματος που θα δώσουμε, είναι καταρχήν μία ευκαιρία να δεσμευτούμε εκ νέου για το 0,7% και να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν θα απέχει πάρα πολύ από τη σημερινή χρονική στιγμή και προς το μέλλον. Τέτοιου είδους δέσμευση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχε δεσμεύσει από τις άλλες αναπτυγμένε χώρες και τι χώρες υψηλού εισοδήματο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι εύκολο. Αν όμω τα αποτελέσματα τη Αντισαμπέμπα είναι πως μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δέσμευση με συγκεκριμένο στόχο, ακόμα και έτσι θα έχουμε κάνει ένα θετικό βήμα. Αλλά θα αποτελέσει και το τέλος της διαδικασίας FFD. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σταθούν με φιλόδοξο και επικοδομητικό τρόπο στην Αντισαμπέβα, στη Νέα Υόρκη. Για μένα δεν πρόκειται για θέμα τακτικής, δεν έχει καν να κάνει με την, επανα... Ε, την εκ νέου δέσμευση και το κατά πόσο αυτή θα ακολουθείται από κάποιες προϋποθέσεις ή όχι, έχει να κάνει με τη στρατηγική προσέγγιση που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά και για το πώς θα αντιμετωπίσει τους αναπτυξιακούς στόχους στο μέλλον. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ανοίξουμε και μία σειρά αποζητήματα ακόμα. Κυρίως σχετικά με το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε και τους εγχώριους πόρους και το θέμα της φορολογίας, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή όχι μόνο όμορφα λόγια και ε, ωραίες προτάσεις, αλλά φιλοδοξία πραγματική. Έτσι ώστε να πετύχουμε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις εφαρμοστικές στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα οποία επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με συγχωρείτε, θα πρέπει να παρακολουθήσετε και τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δίκαιη φορολογία, για την ε, φοροαποφυγή, για τη φοροδιαφυγή, γιατί πολύ σύντομα θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Ήδη έχει γίνει πρώτη συζήτηση μεταξύ επιτρόπων και δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι στην αντισαβέβα εάν δεν έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο εμείς. Οπότε, τα θέματα αυτά της φορολογίας και οι συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά θα επιτευχθούν είτε μέσω αυτού του διακυβερνητικού πάνελ, είτε μέσω κάποιας άλλης μεθόδου και θα αποτελέσουν τμήμα της δικής μας συνεισφοράς στην διαδρομή που θα ακολουθήσουμε ε, κατά τη διάρκεια και μετά τη διάσκεψη της Αντισαμπέβα βεβαίως επαφείται στα κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό θα κάνω όμως προσωπικά ό,τι μπορώ μαζί με τους συναδέλφους μου επιτρόπους έτσι ώστε να είναι αποδεκτά αυτά τα οποία θα προτείνουμε και να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή στόχευση στις ε, μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Uh, uh, και για την όλη διαδικασία και το θεματολόγιο για την ανάπτυξη για μετά το 2015. Αν λοιπόν εξετάσετε την ανακοίνωση θα δείτε πως όντως είναι φιλόδοξη. και πιο πολύ φιλόδοξη από τις προτάσεις που έχουμε και τους δευτάς στόχους της Επιτροπής. Δεν μου αρέσει εγώ να στριμώχνομαι ε, σε άμυνα όταν κανείς συζητά το πόσο φιλόδοξοι είμαστε και η συγκεκριμένη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που θα προς την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και το θεματολόγιο των στόχων δεν θα πρέπει να μας οθεί σε μια αμυντική στάση. Εμείς θα πρέπει τις φιλοδοξίες μας να τις μετατρέψουμε σε μια παγκόσμια ατζέντα η οποία θα ανταποκριθεί στις βασικές εξελίξεις και στις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες που υπάρχουν και στις εταιρικές σχέσεις που αυτές τις στιγμές βρίσκονται ενώπιόν μας όχι μόνο για να διαμορφώσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους σχετικούς στόχους, αλλά για να την εφαρμόσουμε και στην ε, πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτροπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Θα συνεργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είστε σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει κάθε σας προσπάθεια έτσι ώστε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους τους καλεσμένους μας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Και όπως ξέρετε υπάρχει ένα δεύτερο πάνελ με δύο καλεσμένους και θα συνεχίσουμε ευθύ αμέσως. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να κλείσω αυτό το πάνελ ευχαριστώντας για μία ακόμα φορά τους καλεσμένους μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε με το δεύτερο πάνελ. Όπως ανέφερα στην αρχή της ακρόασης, δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει ο Υπουργός Οικονομικών της Αιθιοπίας Ωστόσο, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο έκλεκτους καλεσμένους. Την Κέιλ Χέρλι από την ε, ομάδα του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών που θα μας δώσει τις απόψεις της για το τι θα γίνει μετά το 2015 και έπειτα τον James Jean Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρήσεων και Επενδύσεων. Δεν θέλω όμως να καθυστερήσω άλλο. Θα καλωσορίσω αμέσως την Γκέιλ Χέρλι. από την ομάδα αναπτυξιακών προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ανυπομονούμε λοιπόν να ακούσουμε όσα έχετε να μας πείτε ο, για τις προετοιμασίες του, της διάσκεψης στην Αντίσα Μπέβα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης που με κάλεσε για να μιλήσω σε αυτήν την πολύ σημαντική ακρόαση σήμερα το απόγευμα. Πώς θα πληρώσουμε μετά το 2015. Αυτή είναι μια ερώτηση που αξίζει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ή και εκατομμύρια ή μύρια, μύρια όπως θα έλεγε και το παιδί μου. Πάντως όπως και να έχει τα χρήματα είναι πάρα πολλά και όταν δούμε τα αποτελέσματα της διάσκεψης ε, του Σεπτεμβρίου θα συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι θα μας κοστίσει πολύ. Και θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι καλεσμένοι στο πρώτο πάνελ, ότι δηλαδή το αποτέλεσμα της διάσκεψης της Αντίσα Μπέμπα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η επιτυχία της διάσκεψης θα στείλει ένα μήνυμα πολιτικής στήριξης και δέσμευσης για τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και επίσης θα στείλει ένα μήνυμα και στο, στη Σύνοδο για το κλίμα στο Παρίσι. Είναι λοιπόν μια διάσκεψη η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών κυβερνήσεων. Και η αίσθηση που αποκομίσαμε, όπως και από τον Ταβός, είναι ότι υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπροσωπηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Αντίσα Μπέμπα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω να με βοηθήσετε, να μας βοηθήσετε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό μέχρι την διάσκεψη της Αντίσα Μπέμπα. Προσωπικά έχω παρακολουθήσει στενά τις διαπραγματεύσεις και συμμετείχα στενά σε αυτές και στη Νέα Υόρκη επίσημα και ανεπίσημα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και έχω την εντολή από έξι κράτη-μέλη για να συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε κληθεί να υποστηρίξουμε το έργο των συμμετεχόντων έτσι ώστε να καταφέρουμε να συντάξουμε ένα περιεκτικό κείμενο στο τέλος. Θα ήθελα σήμερα το απόγευμα να εστιάσω σε δύο ε, τομείς. Πρώτα, το πώς θεωρούμε εμείς ε, πώς θα έπρεπε να είναι το έγγραφο που θα προκύψει από την Αντίσα Αμπέμπα, τι θα κάνει τη διαφορά και πού θα, θα βρεθούν τα κονδύλια για να στηρίξουν την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015. Και ε, τα δεδομένου ότι δεν μπορεί να ε, βρίσκεται σήμερα μαζί μας ο Υπουργό Οικονομικών της Αιθιοπίας, θα ήθελα και εγώ να σας εκθέσω τις απόψεις και τις θέσεις που έχουν λάβει ε, διαφορετικές χώρες μέχρι τώρα πού έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε μία συνένεση και πού ε, θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένω προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω μια γενική εικόνα όλου αυτού του κλίματος. Τι κάνει η υπηρεσία μας και τι άποψη έχουμε για τα προβλήματα αυτά. Πρωτό απαντήσω νομίζω πως καλή, καλό θα είναι να κάνω μια σύνοψη της ε, παγκόσμιας προσέγγισης της αναπτυξιακής βοήθειας. Η συμφωνία λοιπόν του Μοντερέι ήταν ένα πραγματικά ρεξικέλευτο κείμενο, διότι περιείχε μια στρατηγική χρηματοδότηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, οι οποίοι είχαν εστιάσει και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η συνένεση του Μοντερέι ανέφερε μεταξύ άλλων τις δεσμεύσεις των ε, κρατών να αυξήσουν το, την κινητοποίηση εγχώριων πόρων και να μειώσουν τη διαφθορά. Καθώς επίσης και να τονώσουν και να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις και σε τοπικό και σε διεθνές ε, επίπεδο. Και όπου υπάρχουν κενά σε αυτέ στη στρατηγική να ε, χρησιμοποιηθούν και να κινητοποιηθούν δημόσιοι πόροι για να καλυφθούν. Να ε, ληφθεί δράση για το χρέος και για ε, την προστασία του περιβάλλοντος. Και οι συζητήσεις και το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων του Μοντερέι είναι πάρα πολύ σχετικό και για την δουλειά μας τώρα και ίσως μάλιστα θα είναι απαραίτητο για να τοποθετηθούμε και να θέσουμε τους στόχους μας για το θεματολόγιο μετά το 2015. Έχουμε μία πολύ περίπλοκη ε, κατάσταση στο χώρο της ανάπτυξης και από την άλλη υπάρχουν εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις στο τι χρειάζεται να γίνει μετά το 2015. Από τη μία έχουμε κληρονομήσει τα παραδοσιακά αναπτυξιακά προβλήματα του παρελθόντος, δηλαδή την ανέχεια, την πείνα, αλλά υπάρχουν και νέα προβλήματα που έχουν προκύψει, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή, η ταχύτατη καταστροφή του περιβάλλοντος και εκεί μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν και οι κυβερνήσεις για να συντονίσουν μια διεθνή δράση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η διεθνής δράση είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τις μεμονωμένε προσπάθειες. Και το θεματολόγιο του 2015 και μετά μας δείχνει πόσο ε, στενά συνδεδεμένοι είναι όλοι αυτοί οι τομεί. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν και ε, και κράτη και εθνικότητες πέρα από αυτά. Καταρχάς, δεν πρέπει να θεωρούμε την ε, ανάπτυξη ως ε, ανεπαρκή, ως περιορισμένη. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν να κάνουν με στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης τις οποίες ακολουθούν οι περισσότερες χώρες και οι οποίες ε, θα συνάδουν με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, η διεθνής βοήθεια συνεχίζει να είναι σημαντική ιδιαίτερα για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, όπως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, πολλές ε, νησιωτικές χώρες. Παίζει λοιπόν, ε, ε λοιπόν ρόλο όχι μόνο στις στοχότερες αλλά και σε πολλές χώρες με μέσο εισόδημα. Το αποτέλεσμα λοιπόν της διάσκεψης της Αντίσα Μπέμπα θα μας δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε μια νέα πνοή ζωής στους στόχους μας και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά την βοήθεια. Επίσης, είναι σαφές ότι οι προκλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν, ιδιαίτερα στη δημόσια χρηματοδότηση, διότι θα χρειαστούν αυξημένοι, αυξημένη δημόσιοι πόροι, ιδιαίτερα σε στην περιβαλλοντική προσαρμογή, στην έρευνα και την ανάπτυξη, την επιστήμη και την καινοτομία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτήν την οικονομική μεταμόρφωση. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς θα διασφαλιστούν οι επαρκείς αυτοί οι πόροι για όλους αυτούς τους τομείς με τρόπο που δεν θα υπονομεύει τους ε, αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Επίσης πιστεύω πως είναι σαφές ότι ε, οι στόχοι για το 2015 και μετά δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από δημόσιους πόρους. Χρειάζονται και εγχώροι πόροι και διεθνείς πηγές και το μεγαλύτερο μέρος των ε, ε, κονδυλίων θα έρθει από ιδιωτικές επενδύσεις, από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας και μέσω της πραγματικής οικονομίας και μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης η φιλανθρωπία και η κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι ε, πολύ σημαντικές και ευπρόσδεκτες. Υπάρχουν κάποιες ε, πάρα πολύ έξυπνες και νοτόμες λύσεις και προτάσεις, όμως δεν είναι αρκετές. Χρειάζεται επίσης και αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές να επενδύσουν στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και τέλος, Ιδιαίτερα στην Ευρώπη αυτή την εποχή είναι σαφές ότι ζούμε σε ιδιαίτερα ασταθείς καιρούς και υπάρχουν πολλοί παράγοντες γι' αυτό. Υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, κλιματική αλλαγή, οικονομικές κρίσεις, σειράξεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο. Και αυτό σημαίνει πως δεν μένει χρόνος για να σκεφτούμε τι θα γίνει με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό τι σημαίνει, ότι η χρηματοδοτική στρατηγική μας πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα ενδεχόμενα των κινδύνων. Και έχουμε πιστεύω τώρα την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο σταθερό πλαίσιο το οποίο θα ε, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις ε, περιπτώσεις κρίσας και θα αποφέρει καρπούς στο απότερο μέλλον. Αυτές ήταν εν ολίγης οι απόψεις μας εν ώψη της διάσκεψης της Αντισαμπέμπα και να σας πω κιόλας ότι αναγράφονται και στο σχετικό νημερωτικό έντυπο καταρχάς χρηματοδότηση, αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή θεωρεί εξίσου σημαντική τη χρηματοδότηση και από δημόσιο και από ιδιωτικό τομέα. Τώρα θα ήθελα να περάσω στο επόμενο στο σκέλος της παρουσίασής μου και να σας ενημερώσω για το καθεστώς των διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα στη Νέα Υόρκη. Καταφέραμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε τις προτάσεις από διάφορες χώρες ή ομάδες χωρών και έχουν ως εξής. Αναπτυξιακή βοήθεια παραμένει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει μία σχετική συνένεση ότι χρειάζεται και δημόσια χρηματοδότηση και παραμένει μάλλον σημαντική η δημόσια χρηματοδότηση. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις, ιδιαίτερα για προγράμματα τα οποία ε, θα χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και υπάρχουν ορισμένες χώρες που τόνισαν ότι οι κίνδυνοι είναι αρκετά υψηλοί για τέτοιου είδους προγράμματα. Επίσης, το πώς θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση και πώς θα υπολογιστεί. Υπάρχουν κάποιες ε, κυρίως νησιωτικές αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες έχουν κάποιες περίπλοκες ε, δομές και έχουν κάνει έκκληση για περισσότερη εκλογήκευση της ε, χρηματοδότησης έτσι ώστε να ε, μπορέσει να χρησιμοποιηθεί καλύτερα στο μέλλον, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, τα κριτήρια που μας βοηθούν για την κατανομή της βοήθειας συζητήθηκαν και συζητήθηκε ιδιαίτερα εάν το κατακεφαλήν εισόδημα είναι αρκετό ή κατάλληλο για να μας ε, κάνει να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το αν χρειάζεται ε, μια χώρα αναπτυξιακή βοήθεια ή όχι. Επίσης, ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις για την ε, φορολόγηση, συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα και τις παράνομες ροές κεφαλαίου. Ιδιαίτερα α, τόνισαν κάποιες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνες και έχουμε δει πρόοδο στην διεθνή συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα, πρέπει να πω. Έχουμε δει την πρόοδο αυτή στα αφορά του G20 για παράδειγμα. Και θεωρούμε πως θα έπρεπε να αφιερωθεί ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό φόρουμ για αυτές τις συζητήσεις έτσι ώστε να προωθηθούν αλλαγές. Επίσης, οι ίσοι κανόνες του εμπορικού ανταγωνισμού, ανάπτυξη των υποδομών, είναι εξίσου σημαντικά. Και πέραν αυτών πιστεύω πως υπάρχει μια γενική παραδοχή ε, για το ότι χρειάζεται ένας καινούριο ε, μηχανισμός που θα μας βοηθά να αξιολογούμε την επιτυχία κάθε προγράμματος. Χρειάζεται λοιπόν ένας ολοκληρωμένος εποπτικός μηχανισμός. Έγιναν κάποιες προτάσεις για να χτίσουμε πάνω σε υπάρχουσες δομές αλλά και κάποιες χώρες ε, πρότειναν πολύ πιο φιλόδοξα προγράμματα που θα μετρούν και τις ε, στατιστικές δυνατότητες καταμέτρησης. Επίσης, όσον αφορά τη δομή του εγγράφου εργασίας, να σας πω ότι Υπάρχουν ορισμένε απόψει που υποστηρίζουν πως πρέπει να κρατήσουμε τη δομή του εγγράφου του Μοντερέ και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες υποστηρίζουν ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια τελείω διαφορετική ε, δομή βασισμένη σε δουλειά εμπειρογνωμόνων. Τα προσχέδια με τα οποία εργαζόμαστε τώρα έχουν ως άξονά τους ε, κεφάλαια για κινητοποίηση ιδιωτικών ε, κεφαλαίων για διεθνή οικονομική συνεργασία, συστημικά ζητήματα. Υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο για την καινοτομία και την τεχνολογία. Και επίσης ένα κεφάλαιο για, το, για την παρακολούθηση του FFT. Θα σταματήσω εδώ. Παραγματικά αναφέρθηκα μόνο επιφανειακά στα ζητήματα της ε, αναπτυξιακής χρηματοδότησης και πιστέψτε με είναι τεράστιο το θέμα με πολλές παραμέτρους. Αλλά θέλω να συνεχίσουμε την ε, συζήτηση. Μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα ακόμα, για την ε, διεθνή συνεργασία και αν θέλετε μπορώ να απαντήσω με περισσότερες λεπτομέρειες με τη μορφή σχολείου. Και θα ήθελα να κλείσω με κάτι θετικό. Θα ήθελα να πω ότι όλοι έχουμε ευθύνη, συλλογική ευθύνη για την επιτυχία ε, του προγράμματος αυτού και πιστεύω πως έχουμε τη δυνατότητα να οδηγηθούμε σε κάτι ε, πολύ καλύτερο από το έγγραφο του Μοντερέι, διότι έχουμε τις ε, δυνατότητες και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογία ε, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τις οποίες δεν είχαμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω πως εάν καταφέρουμε να έχουμε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη θα έχουμε μεγάλο όφελος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ειδικά από εσά που είσαστε στο επίκεντρο των, της προετοιμασίας για την Αντισαμπέμπα. Είδαμε πώς βλέπουν το πράγμα οι, τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα θα συνεχίσουμε. Θα παραμείνουμε στην ευρύτερη οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο James Zan. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που ε, συμμετέχω σε αυτό το πολύ σημαντικό φόρουμ και που μπορώ να ε, συμβάλλω σε αυτή την σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Ο ρόλος μας ε, σε αυτή τη φάση είναι να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο ε, input και προώθηση σε αυτό το σύνολο των τριών ε, διασκέψεων και στην Αντισαμπέμπα και μετά στη Νέα Υόρκη αλλά και ε, στο Παρίσι για την κλιματική αλλαγή. Εμείς έχουμε προετοιμάσει ήδη πέρσι μία σχετική έκθεση υπό το ε, ε, ε, σχέδιο δράσης για την επίτευξη βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Τώρα, η ανάγνωση μπορεί να είναι ποσοτική. Τι χρειάζεται, τι ποσότητες χρειάζονται για μια τέτοια βιώσιμη ανάπτυξη και δεύτερη διαδρομή, ας πούμε, σκέψης είναι το πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Αυτό το μονοπάτι θα ακολουθήσω και στην παρουσίασή μου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα σας δώσω ε, ε, το, μία εικόνα των πολλών και διαφορετικών σημαντικών παικτών που ε, σχηματίζουν το περιβάλλον της ε, της χρηματοδότησης θα ήθελα να πω ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης δεν είναι μια απλή χρηματοδότηση, δεν είναι απλή χρήση χρημάτων δηλαδή και κονδυλίων. Ε, βασικά ε, το, το κύριο θέμα είναι η κινητοποίηση των ε, πόρων μετά η μεταστροφή τους σε κονδύλια και όταν τα χρήματα μαζεύονται να γίνονται επενδύσεις με τρόπο ώστε ε, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι να ελαχιστοποιηθούν και το ε, αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί. Οι κίνδυνοι είναι συγκεκριμένοι. Τους, ο Τζέσε τους ε, έχει αναπτύξει. Αυτό που θέλουμε εδώ είναι μία σειρά δράσεων. Επομένως ένα συνολικό σχέδιο δράσης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την κινητοποίηση των πόρων, την πρόθεσή τους προς κρίσιμους τομείς υποδομών όπως είναι ας πούμε ε, έργα για την πρόσβαση στο νερό κτλ και μετά ε, να, αυτό που είπα προηγουμένως, να υλοστοχιοποιηθούν οι κίνδυνοι και να, ε, να ε, έχουμε όσο γίνεται πιο μεγιστοποιημένο αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί μας αναφέρονται στην περίοδο 15 με 30 το συνολικό ε, ποσό θα μπορούσε να είναι περίπου 3,93 εκατομμύρια ε, ε, δολάρια για τις αναπτυσσόμενες χώρες. αυτά τα 3,93 ε, για αυτά τα δολάρια, για αυτά τα ε, χρήματα βλέπουμε ότι ε, παρόλα αυτά θα υπάρξει ένα ετήσιο χάσμα περίπου 2,5-3 για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι ένα τεράστιο χάσμα που δεν μπορεί να, τον, ε, ε, να το καλύψει ο δημόσιος τομέας. Άρα χρειαζόμαστε ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Βεβαίως είναι θεμελιώδους σημασίας η δημόσια επένδυση, αλλά και η ιδιωτική επένδυση είναι απαραίτητη. είδαμε ε, από κοντά όλους τους τομείς έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι τομείς ε, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερα και ποιοι λιγότερα. Ποιοι είναι οι τομείς ε, οι οποίοι απαιτούν ή χρειάζονται περισσότερη ιδιωτική επένδυση και αντίστοιχα ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο δημόσια επένδυση. Στην ουσία σε τομείς όπως ας πούμε οι υποδομές ή όπως η επισητιστική ασφάλεια, βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις ιδιωτικού τομέα, ενώ ε, στην εκπαίδευση, ας πούμε, μπορεί να παίξει περισσότερο ρόλο η δημόσια εκπαιδευση πουμε μπορει να παιξει περισσοτερο ρολο η δημοσια επενδυση Είδαμε τώρα ε, και μελετήσαμε τους διαθέσιμους πόρους. Ε, βεβαίως όλοι οι ε, ε, συνολικότεροι πόροι, όλα τα assets δεν μπορούν να επενδυθούν άμεσα και δεν είναι εύκολο ε, να πούμε ότι 5 ή 10% των assets θα χρησιμοποιηθούν ε, άμεσα Ξέρουμε ότι σε ορισμένες περιοχές μάλιστα και σε ορισμένες χώρες αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο, κυρίως σε χώρες με πολύ χαμηλό εισόδημα. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν ας πούμε πολλές ε, φιλανθρωπικές ε, ε, οργανώσεις οι οποίες δρούν επιτόπου και είναι χώρες στις οποίες δεν πηγαίνουν συχνά οι επενδυτές γιατί η επιστροφή της επένδυσης είναι πολύ χαμηλή ή πολύ δύσκολη ή επίσης ε, είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλή ικανότητα διαχείρισης ε, των προγραμμάτων. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και το πρόβλημα της έλλειψης τεχνογνωσίας, πραγματογνωμοσύνης, ακόμα και για τις ε, επενδύσεις. Ε, τα pipeline projects τα οποία είναι έτοιμα ε, για την επενδυτική τους φάση σε μερικές περιοχές είναι πάρα πολύ, λίγες, πάρα πολύ λίγα και επομένως τη θέση ε, της επένδυσης παίρνουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε επένδυση στους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους μέσω ε, προγράμματος δράσης ε, που θα βελτιστοποιήσει και θα πολλαπλασιάσει το αποτέλεσμα τους. χρειαζόμαστε ε, δέσμοι ε, μέτρων. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θέλουμε οπωσδήποτε ε, να αναφερθούν στην διάσκεψη για την αναπτυξιακή, για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και μάλιστα να υποστηρίζεται η άποψη αυτή από συγκεκριμένα έγγραφα. Πρώτα απ' όλα, Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά ε, θεσμών και ε, ε, εργαλείων προώθησης των στρατηγικών. Στις περισσότερες χώρες, τουλάχιστον στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουμε εταιρείες αναπτυξιακές ή εταιρείες προώθησης της ανάπτυξης. Όμως, οι εταιρείες αυτές συνήθως δεν έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν προγράμματα τουλάχιστον στον τομέα της ε, βιώσιμη, των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Ε, ε, άρα έλλειψη τεχνογνωσίας, έλλειψη δομών και υποδομών. Άρα αυτό που θέλουμε είναι όλες αυτές οι επενδυτικές υπηρεσίες να γίνουν ε, το, μέσο ε, το οποίο θα αναπτύξει τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους μέσα από την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας. Τρίτον, ε, στην, στο Διεθνές Επενδυτικό Καθεστώς βλέπουμε ότι ακολουθείται το, το, μοντέλο, το πρότυπο των πολυμερών συμφωνών, αλλά δεν Υπάρχει όμως ε, πολυμερές ε, σύστημα το οποίο να αναφέρεται στην χάρτα του 94. Μια και δεν υπάρχει ε, πολυμερές καθεστώς επενδύσεων, Ε, έχουμε διμερείς ε, ή μερικές συμφωνίες ε, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πληθώρα πάνω από 3.200 τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες, κατακαιρματισμό επομένως μεγάλο, πολυγλωσία που δυσκολεύει την κατάσταση. Μελετώντας δε αυτές τις ε, συμφωνίες ε, διαπιστώνουμε ότι είναι εξαιρετικά ελλειπές το αναπτυξιακό ε, υπόβαθρο με διαρθρωμένο τρόπο βέβαια. Άρα αυτή τη διάσταση πρέπει να τη δουλέψουμε. Επίσης ε, είναι ε, πολύ διαταραγμένη η ισορροπία ε, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επενδυτών. Και αυτή είναι η δεύτερη δράση που πρέπει να αναλάβουμε στα πλαίσια της διάσκεψης της Αντισαμπέμπα και οπωσδήποτε θα πρέπει να μπει και στα έγγραφα. Τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε νέο προσανατολισμό των κινήτρων της επένδυσης. Εάν ε, δει κανεί τα επενδυτικά προγράμματα σε πάνω από 120 χώρες, διαπιστώνει ότι η κινητροδότηση που έχει δοθεί σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες ε, είχαν στόχο την ανάπτυξη της ε, τοπικής ε, αποτελεσματικότητας και την αύξηση της ελκτικότητας που μπορούν να έχουν οι χώρες αυτές. Αλλά έχουν παραμεληθεί ουσιαστικοί τομείς όπως είναι οι υποδομές στην επισητιστική ασφάλεια, στην πρόσβαση στο νερό, στην εκπαίδευση, στην υγεία κτλ στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα πρέπει να καλυφθεί ε, αυτό το χάσμα. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να η εστίαση να γίνει προς βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους μέσα από την καθαρή στοχοθέτηση και κινητροδότηση των εταιριών. Επομένως, ε, πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ε, καθολικά που να αφορούν την κινητροδότηση. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένα καλό σύστημα εγγύησης των, ε, και διασφάλισης των επενδύσεων. Μια άλλη σειρά δράσης ε, αφορά τους τοπικούς βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Ξέρουμε ότι υπάρχει το ζήτημα της ε, οικονομίας κλίμακος. Χρειαζόμαστε μεγάλα προγράμματα, mega projects, μεγάλες ε, διαρθρωτικές επενδύσεις, συγγνώμη, επενδύσεις σε υποδομές έτσι ώστε ε, μία ομάδα χωρών από κοινού ε, να ε, αποτελέσουν θελκτικό στόχο και προορισμό για μία μεγάλη επένδυση. Ε, να δημιουργηθούν επίσης τοπικές, ε, ε, τοπικές ομάδες, τοπικές συνενώσεις, clusters, έτσι ώστε να υπάρξει μία προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά. Επομένως, ε, βιομηχανικά κλάστερς, ε, ε, δημιουργία κεντρικών πόλων έλξης σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, όσον αφορά τις εταιρικές σχέσεις, έχουμε δει ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν ε, οι υπηρεσίες προώθησης και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την εξέβρεση αναπτυξιακών ε, ε, ή επενδυτικών εταίρων, αλλά Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό, κυρίως για τις λιγότερο αναπτυχημένες χώρες, είναι να προχωρήσουν εταιρικέ σχέσεις, έστω και αν δεν είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για, τις, για τους επενδυτές, να αλλάξει η δομή των επενδύσεων, έτσι ώστε μέσω τριμερούς χρηματοδότησης να μπορέσουν να προωθηθούν κάποια ιδιαίτερα κεντρική σημασίας προγράμματα. Γνωρίζουμε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές αυτή τη στιγμή ε, ε, ε, είναι, αποτελούν πεδίο τεράστιων μετακινήσεων πόρων και τεράστιων ροών. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ε, ροές αυτές, να χρησιμοποιήσουμε σωστά ε, τα κίνητρα τα οποία μπορούν να δοθούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα έτσι ώστε να τον ενθαρρύνουμε τον τομέα αυτό να, να ενδιαφερθεί για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Το Κυριότερο βεβαίω είναι να αλλάξουμε την επιχειρηματική νοοτροπία. Η νοοτροπία του επιχειρήν θα πρέπει ε, ε, να ξεκινήσει να αλλάζει ήδη από τα πανεπιστήμια, από τα ε, business schools. Κοιτάξτε, η κλασική θεωρία είναι πριν κάνεις μια επένδυση να δεις το μέγεθος της αγοράς, τις δυνατότητες της αγοράς, την, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επένδυσης ε, και έτσι ε, ε, προωθείται η επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά επιχειρηματιών, να ανοίξουμε νέες οδούς δυνατοτήτων επένδυσης σε άλλες χώρες όπου μπορούν να εξευρεθούν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας ε, ε, μέσα από ένα επιχειρήν πιο ε, υπεύθυνο. Αυτά ήθελα να σας πω. Είχα και άλλα πολλά να σας πω, αλλά βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε, αλλά έχουμε και πάρα πολλές ιδέες τις οποίες θέλουμε να σας μεταφέρουμε ε, και εάν εφαρμοστούν οι ιδέες αυτές ε, είμαστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις ε, θα γίνουν σωστά, θα γίνουν σε κεντρική σημασία τομείς και οπωσδήποτε θα παράξουν μεγάλο και πολλαπλασιασμένο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I'm going to give the floor now. You have the floor. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ερωτήσεις έχουμε. Ευχαριστώ πολύ η αναφορά που έγινε στο ότι οποιαδήποτε βοήθεια απαιτεί έναν εταίρο, έναν ομόλογο, μία υπευθυνότητα από την άλλη πλευρά, δυστυχώς έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Όταν ταξιδεύει κάποιο στην τρίτο κόσμο, και κυρίω στην Αφρική αλλά και αλλού το ίδιο συμβαίνει, αντιμετωπίζουμε το εξή. Χιλιάδες έργα που έχουν υλοποιηθεί, που αποτελούν απλώς κενά ε, και, ε, και λυφή κενά, ε, που δεν υπάρχουν. Σχολεία δηλαδή που χτίστηκαν αλλά έμειναν κτίριο. Νοσοκομεία που χτίστηκαν με διεθνή βοήθεια που δεν υπάρχουν φάρμακα για γιατροί. Άρα λοιπόν οι δεσμεύσει των ε, τοπικών κυβερνήσεων που είναι η διαχείριση, η συνδιαχείριση ε, αυτών των υποδομών, δηλαδή δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, δεν γίνεται στην πράξη στην πράξη. Δεν στέλνουν γιατρούς, δεν στέλνουν καθηγητές, δεν τους πληρώνουν και έτσι έχουμε κενά κτίρια με μια πινακίδα έξω από το κτίριο που λέει χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΗΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να υπάρχει τίποτα πίσω από αυτή την πινακίδα. Και αυτό συνέχεια. Έχει νόημα να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε έργα για τα οποία έχουμε και την εμπειρία και την αίσθηση πως τελικά θα καταλήξουν σε άδεια κτίρια σε εγκαταστάσεις που έχουν λαιλατηθεί γιατί οι κυβερνήσεις που μας ζητάνε βοήθεια δεν έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις τους να διατηρήσουν και να συντηρήσουν και να συμμετάσχουν στη διαχείριση με, τα, ε, με τις πόρους που έχουν σύμφωνα και με τα όσα έχουν υπογράψει. Άρα λοιπόν τι νόημα έχει να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε νέα project και θα το πω με κάθε ειλικρίνεια που αποτελούν απλώς οχήματα διαφθοράς γιατί αυτές οι οικοδομές και αυτές οι κατασκευασίες εργασίες αναλαμβάνονται σε κάποιον. Όχι τυχαία, σε κάποιον που έχει σχέση με την κυβέρνηση. Με κάποιον από την κυβέρνηση, με κάποιον από το δημόσιο, από το κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά εμεί χρηματοδοτούμε υποδομές που θα μείνουν άδειε μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, θα τι εγκαινιάσουν, θα βγάλουν φωτογραφίε, θα δείξουν τα παιδιά, θα δείξουν του αρρώστου, θα δείξουν του γιατρού. Και θα σα πω κάτι που είναι αρκετά συνηθισμένο. Ότι είναι σαν να βλέπει κανεί ε, κάποια παράσταση ε, όπω έκανε ο γνωστό ε, Ποτέμκιν. Ε, Παραστάσει φαντάσματα, εγκαταστάσει φαντάσματα με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει νόημα και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Αντί να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδου έργα με κυβερνήσεις που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους, πριν από την επόμενη χρηματοδότηση να του ζητήσουμε να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν όσα έχουν ήδη υπογράψει. Διαφορετικά καμία νέα χρηματοδότηση. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι εμείς να εγκαινιάζουμε κτίρια, αλλά να λειτουργούν τα κτίρια αυτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. για τις επενδύσεις και πολύ με ενδιαφέρει η ιδέα αυτή που παρουσιάσατε που ζητά να εξασφαλίζουμε πως οι αναπτυσσόμενε χώρες να κερδίσουν περισσότερα από τις επενδύσεις όταν οι ίδιες επενδύουν στη χώρα τους. Εγώ στην προηγούμενή μου ζωή εργαζόμουν για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια και πολλές φορές ε, η ερώτηση από την τοπική κυβέρνηση είναι ντόπιοι τι θα κερδίσουν. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε επιχειρήσεις από τη δική μας Ήπειρο που πάνε στις χώρες αυτές και παρόλα αυτά δεν συμμορφώνονται με κανέναν κανόνα είτε σε σχέση με το περιβάλλον, Και πώς μπορούμε να υποχρεώσουμε τις εταιρείες αυτές να γίνουν καλύτερες. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις χώρες έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν με τους επενδυτές. Πώς διαπραγματεύεσαι με έναν επενδυτή. Δηλαδή το κέρδος του σχεδιασμού υπάρχει. Στην έκθεσή σας πέρσι, όπου μιλήσαμε για την επένδυσή στην Αφρική και κάποιες από τις αναδυόμενες οικονομίες αναρωτήθηκα πώς αντιμετωπίζετε εσείς την κατάσταση ασφάλειας και το πώς επηρεάζει αυτό τις επενδύσεις και την εμπιστοσύνη. Γιατί τελικά σήμερα δεν το συζητήσαμε αυτό. Ζούμε δηλαδή σε έναν κόσμο, γιατί το είπε χτες ο Επίτροπος, ότι χωρί ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχουν τεράστιε προκλήσει για την ασφάλεια στι χώρε Αφρική. Η Μπόκο Χαράμ, για παράδειγμα, ε, ακραίες οργανώσεις που στοχοποιούν και προσπαθούν να ε, δημιουργήσουν συνθήκες αστάθειας. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Δηλαδή επένδυση στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς που θα είναι οι νέοι επιχειρηματίες που θα ε, επενδύσουν στις φτωχές χώρες. Τι γίνεται αν αυτές οι φτωχές χώρες έχουν παράλληλα και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικής ανασφάλειας ή αστάθειας. Έχετε το λόγο. Είμαι ο James Bartholomew από τη Γενική Γραμματεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τον James Χιάν έχω ένα θέμα. Μιλήσατε για το πολυμερές παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε για παράδειγμα για ένα επενδυτικό καθεστώς που θα ακολουθεί τους κανόνες ε, του Δουνουτού ή του ΠΟΕ. Αλλά δεδομένου του τέλματος που διαπιστώνει κανείς στις διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ τα τελευταία χρόνια και των κρίσεων σε επίπεδο παγκόσμιας ασφάλειας, πιστεύετε πως υπάρχει οποιαδήποτε όρεξη για ένα ακόμα πολυμερές όργανο. Και πώς μπορούμε να ε, εξάψουμε την περιέργεια και των υπολείπων κρατών ε, στον κόσμο, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα για κάτι τέτοιο. Έχω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, έχει να κάνει με το αφήγημα που θα χρησιμοποιήσουμε. Uh, challenges, but, um... Νέες προκλήσεις. Νέα αφήγηση. Αποτελούν όλα αυτά φυλασικής. Γιατί πια λένε πως η επίσημη αναπλεξική βοήθεια δεν είναι πια τόσο σημαντική. Μα γιατί, επειδή ακριβώς είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε τους συγκεκριμένους στόχους, Σε ποιο βαθμό λοιπόν αντιμετωπίζουμε δικαιολογίες και προφάσεις. Γιατί για τα υπόλοιπα, για τους εγχώριους πόρους, για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, όλα αυτά είναι ήδη ε, στην ατζέντα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δεύτερο ερώτημα, σε σχέση με την διαδικασία προετοιμασίας για την διάσκεψη της Αντισαμπέπα. Τι να περιμένουμε. Ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις που θα πάρθουν. Ο Τζέιμς αναφέρθηκε σε μια νέα προσέγγιση και μια νέα καθοδήγηση των όσων σκοπό να επενδύσουν. Τι προετοιμάζετε αυτή τη στιγμή εσείς, τι περιμένουμε για το άμεσο μέλλον. Μια νέα κατεύθυνση στις επενδυτικές προσπάθειες. Είναι αυτό το μέσο για να εξασφαλίσουμε πως είναι πιο βιώσιμη η ιδιωτική επένδυση και βοηθά στην ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποιοι πιο βιώσιμοι στόχοι. Φόροι. Επίκυνται κάποιες πολιτικές αποφάσεις για τη φορολογία, για, τις, για τη φορολογία των ε, διεθνών επιχειρήσεων, ε, διεθνή φορολόγηση κερδών στην Αντισαμπέβα, κάτι αντίστοιχο. Και τέλος, Γκέιλ. Ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι προτείνεται. Τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα πρέπει να είναι η δική μας συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη την γενικότερη διάθεση ε, στην ομάδα προετοιμασίας. Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα ήταν χρήσιμο από πλευράς μας για να είναι επιτυχής η διάσκεψη στην Αντισαπέμπα. James, να απαντήσεις πρώτος? Thank you very um, uh, Για το πρώτο σχόλιο, για την βοήθεια και την αποδοτικότητα της βοήθειας και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει, το πιο σημαντικό που θίξατε είναι η βιωσιμότητα των έργων αυτών. Το πρόβλημα εκπορεύεται από τρεις πηγές. Πρώτα απ' όλα, αυτού του είδους τα έργων βοήθειας ακολουθούν μία κατακαιρματισμένη προσέγγιση, οπότε δεν είναι κομμάτι ενός πακέτου για εκείνη την περιφέρεια, για εκείνη τη χώρα, για εκείνο τον κλάδο. Δεύτερον, δεν έχουμε αρκετές βιο... Ε, μελέτες βιωσιμότητας ε, πριν ξεκινήσουμε. Και τρίτον, διακυβέρνηση. Καλή διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση και διαχείριση έργων από την ίδια τη χώρα. Ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε και βρίσκεται στην εκθέσή μας είναι όταν προσφέρουμε τέτοιου είδους βοήθεια και όταν ε, προσελκύουμε επενδύσεις θα πρέπει σε επίπεδο πολιτικής χάραξης να τοποθετούμε και κάποιους δείκτες που θα επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ποια θα είναι τα εργαλεία παρακολούθησης, έτσι ώστε να πούμε τι ακριβώς είναι ε, βιώσιμο έργο. Ποια έργα θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε κάποιους δείκτες αποδοτικότητας, κάποιους δείκτες παρακολούθησης και βεβαίως ε, τους μηχανισμούς αναφοράς. Και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών και άλλους ε, παίκτες έτσι ώστε να παρακολουθούν και να επιτηρούν και ήδη το έργο. Έχουμε ένα πακέτο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχουμε και την πρωτοβουλία που λέγεται βιώσιμα ε, χρηματιστήρια οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως παραδείγματα. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε το συντονισμό που έχουμε μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Στην έκθεση μας εμείς αναφερόμαστε σε ένα είδος ομίλου που θα είναι ένας μηχανισμός συντονισμού όλων των πολυμερών οργανώσεων και τραπεζών έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν το θέμα της βιωσιμότητας κάποιου επενδυτικού έργου ή κάποιου αναπτυξιακού έργου. Άρα λοιπόν να έχουμε ε, μια τέτοιου πολύ ε, μερή προσέγγιση. Σχετικά τώρα με τι επενδύσει και την ασφάλεια, όντω αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Βεβαίως, ε, το θέμα είναι ε, ποιο έκανε το αυγό ή την κότα. Γιατί χωρίς επενδύσεις δεν έχει κανείς βιώσιμη ειρήνη, αλλά χρειάζεται και ειρήνη για να προσελκύσει τις επενδύσει. Άρα λοιπόν είναι αλληλένδετα. Η κοινότητα των δωρητών θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μεταξυραξιακές χώρες, ώστε να προσελκυθούν εκεί οι επενδύσεις και η ανάπτυξη και να διευκολυνθεί η βιώσιμη ειρήνευση εκείνης της περιοχής. Δεν νομίζω όμως πως οι επενδυτές θα πάνε σε ανασφάλεις περιοχές για να επενδύσουν. Αυτό είναι το δίδυμα της πραγματικότητας τώρα για το πλαίσιο της πολυμερούς ε, επένδυσης να γίνω πιο σαφής. Εμείς δεν είμαστε υπέρ ενός πολυμερούς πλαισίου για επενδύσεις, πολυμερούς επενδυτικού πλαισίου αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε και εσείς δεν υπάρχει καμία όρεξη για κάτι καινούριο ακόμα. Αυτό το οποίο προκρίνουμε είναι ελήψη ενός πολυμερούς πλαισίου για τις επενδύσεις να χρησιμοποιούμε τις ε, υπάρχουσες συνθήκες για τις επενδύσεις. 3.600 κάτι αυτή τη στιγμή. Έχουν συγγραφεί, έχουν υπογραφεί πριν από 20, 30, ακόμα και 10 χρόνια. Δηλαδή, σε δεκαετία του 70, του 80 και όλες αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν τη διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή, ακολουθούσαν το παλιό μαντελό και όχι το καινούριο με τις νέες στρατηγικές ανάπτυξης. Γι' αυτά, σε αυτά πρέπει να στραφούμε και να αναθεωρήσουμε αυτό το καθεστώς, έτσι ώστε να εξυγχρονίσουμε τις υφιστάμενες συνθήκες και να εξασφαλίσουμε πως οι 40 συνθήκες που αυτές τις στιγμές βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ 90 χωρών να ε, προχωρήσουν. Ξέρουμε πως κάθε δεύτερη εβδομάδα υπογράφεται μια νέα επενδυτική συνθήκη και πρέπει να πω πως Εκεί πρέπει να δράσουμε και να εξασφαλίσουμε που συνέσαι αυτές οι συνθήκες όντω εξυπηρετούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτός είναι ο στόχο μα. Προς τα εκεί κινούμεθα και είμαστε υπέρ μια αναθεώρησης εκεί. Υπάρχει ευρεία συνένεση πω χρειάζεται αυτή. Οπότε από αύριο στην Γενέβη θα έχουμε άτομα πάνω, πάνω από 100 συνέδρους για να συζητήσουμε πώς μπορούμε αυτή την ε, συνθήκη να την αναθεωρήσουμε, την Άγκαρ. Και πρέπει να σας πω πως για την τελευταία σας ερώτηση για το κατά πόσο ε, υπάρχουν δύο διαδρομές που ακολουθούμε και αν θα λειτουργήσουν, ε, προσπαθώ να σας πω πως καταρχήν στο έγγραφο για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών για ε, τη στρατηγική για αυτές τις χώρες, δηλαδή προσπαθούμε να εντάξουμε αυτά τα στοιχεία, να υπάρχουν τα πορίσματα αυτά στην τελική μορφή, έτσι ώστε όταν συνεδριάσει η ομάδα εργασίας για τους στόχους και για τα εργαλεία να τα έχουν, και το δεύτερο είναι πως και εμείς στη δική μας οργάνωση έχουμε την δική μας εντολή, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι, ε, να παρακολουθούμε τις επενδύσεις για να δούμε πώς οι μεμονωμένες χώρες ε, εκτελούν ε, αυτές τις υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χέρλη θα απαντήσει τώρα στις ερωτήσεις. Μάλιστα μου δίνετε την ευθύνη να συνοψίσω και να ολοκληρώσω. Εξαιρετικές οι ερωτήσεις σας, καταρχάς, θα ήθελα να πω. Ε, και τώρα όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για την αποτελεσματικότητα ε, και για τα χιλιάδες παραδείγματα αποτυχίας. Πραγματικά, ε, δεν τίθεται θέμα. Έχουν αποτύχει και έργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί με δημόσια κονδύλια. Αλλά φυσικά υπάρχουν και χιλιάδες παραδείγματα όπου είχαμε δει μεγάλη επιτυχία και πραγματικά ε, αυτά τα έργα έκαναν τη διαφορά και άλλαξαν τις ζωές των ε, ανθρώπων. Πιστεύω πως έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια και Τώρα πλέον είμαστε περισσότερο, από, περισσότερο προσανατολισμένοι στην ανάληψη ευθύνη, στην ε, συμμετοχή των ε, δωρητών, στον καθορισμό προτεραιοτήτων, στην δημιουργία τοπικών θεσμών, σε όλα αυτά που έχει εμπειρία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω πως έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και Ελπίζω να τονιστεί αυτή η πρόοδος στο έγγραφο που θα παραδώσουμε στη διάσκεψη της Αντισαμπέμπα. Τώρα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ακραία φτώχεια θα συγκεντρωθεί στα ευάλωτα κράτη τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Και εκεί έχουμε και τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Θα είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα προς επίλυση για τη διεθνή κοινότητα και πραγματικά χρειάζεται κοινή δέσμευση και κοινή συνεργασία, μακροπρόθεσμα. Τώρα, το νέο σχέδιο, το νέο πρόγραμμα και αν αυτό είναι δικαιολογία, αν υπάρχουν δισταγμοί για να αναλυφθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Να σας πω ότι στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων αυτό που μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον ήταν το πόση έμφαση έδωσαν οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, στο ρόλο των δημόσιων οικονομικών και πόσο αντίθετες ήταν με αυτό οι ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες στήριζαν τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Η έμφαση λοιπόν είχε δοθεί στους ε, δημόσιους ε, πόρους και αυτό είναι και, και μια σημαντική ένδειξη των προτεραιοτήτων της κάθε χώρας. Πολλές ανεπτυγμένες χώρες Αντίθετα, τόνισαν ότι η κινητήρια δύναμη είναι ένας δυνατός ιδιωτικός τομέας που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και εμείς τώρα για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τους ιδιωτικούς με τους δημόσιους πόρους και να χρησιμοποιήσουμε αποδοτικότερα τα λιγοστά κονδύλια που διαθέτουμε πρέπει να αναγνωρίσουμε μεν ότι υπάρχουν αυτές οι εντάσεις και αυτές οι διαφορές, αλλά από την άλλη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε είδους χρηματοδότηση είναι εξίσου σημαντική και έχει το δικό της ρόλο στην αναπτυξιακή βοήθεια κάποιες μορφές χρηματοδότησης είναι για παράδειγμα κατάλληλες για συγκεκριμένα κράτη, για συγκεκριμένα έργα. Και τέλος, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μπορούμε να περιμένουμε από εκείνη. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα έγγραφο που δείχνει τις προοπτικές μας και με τα χαράς να το μοιραστώ μαζί σας τις προοπτικές μας και υπάρχουν κάποιες προτάσεις από τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με το ποιοι τομείς είναι πιο σημαντικοί για την ε, χρηματοδότηση μετά το 2015. Υπάρχουν δεσμεύσεις και για ποσότητα και για ποιότητα και πιστεύω πως ε, έτσι θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για το τι θα γίνει μετά το 2015 και για το ποιους στόχους πρέπει να θέσουμε. Μία από τις ε, προτάσεις μας για καλύτερη επιλογή είναι να μην χρησιμοποιούμε το κατακεφαλήν εισόδημα ως ε, πλοηγό, αλλά να χρησιμοποιούμε και άλλους δείκτες σε συνδυασμό με το κατακεφαλή εισόδημα, όπως για παράδειγμα την κλιματική αλλαγή, την ε, ευαισθησία στην κλιματική αλλαγή, το, το μέγεθος του χρέους μιας χώρας που εξαρτάται από εξωτερική χρηματοδότηση, εάν συμπεριληφθούν και αυτά, πιστεύω πως θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης και έτσι να στοχεύσουμε την κατανομή των πόρων καλύτερα. Θα συνεχίσουμε φυσικά να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, αλλά στο τελευταίο έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών τονίστηκε η ανάγκη να διερευνήσουμε τη σχέση δημόσιας και ιδιωτικής ε, χρηματοδότησης και να δούμε πόσο μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο για την καλύτερη χρήση αυτών. Τώρα, τι βήματα χρειάζεται να πάρουν οι χώρες έτσι ώστε να μπορέσουν να κατευθύνουν την, ε, το ιδιωτικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή βοήθεια. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να τιμολογήσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα μπορούσαμε να καταστήσουμε υποχρεωτικούς μερικούς ε, μέχρι τώρα προαιρετικούς ε, κανόνες, όπως για παράδειγμα εκθέσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Και τέλος, να απαντήσω για το χρέος, αν και δεν το ανέφερε στην παρουσίασή μου. Ο Τζέσι ανέφερε το χρέος ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα δεν θα αναλύσω τα υπέρ και τα κατά ενός ε, πολυμερούς διεθνούς πλαισίου για να αναδιάρθρωση χρέους, αλλά θα περιοριστώ στο να πω ότι κάποιες χώρες αποκλείστηκαν από την πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες. Και αυτή η πρωτοβουλία πραγματικά βοήθησε στο να μπουν σε μια θετική πορεία ανάπτυξης αυτές οι πάρα πολύ φτωχές χώρες. Και αυτές οι χώρες που αποκλείστηκαν είναι κατά κύριο λόγο μικρές νησιωτικές χώρες που παλεύουν με υπέρογκο χρέος. Και πιστεύω πως πρέπει να δούμε τι διδάγματα αντλήσαμε από το παρελθόν και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τις χώρες που είναι τώρα υπερχρεωμένες. Και να δούμε πώς μπορούμε να γίνει το χρέος βιώσιμο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους καλεσμένους στο δεύτερο πάνελ, αλλά και όλους εσάς δεν θα κάνω κάποια συμπερασματικά σχόλια. Πιστεύω να συμμερίζεστε κι εσείς την άποψή μου ότι είχαμε μία ιδιαίτερα χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και πιστεύω πως συνειδητοποιούμε όλοι ότι μία ισχυρή συνεργασία χρειάζεται διάλογο. Χρειάζεται ισχυρό διάλογο όχι μόνο μεταξύ των θεσμικών οργανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε διεθνές επίπεδο με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με άλλους διεθνείς οργανισμούς έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα επιτυχημένο ε, αποτέλεσμα στη διάσκεψη της Αντισαμπέμπα. Χρειάζεται πίεση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αυτόν τον ηγετικό ρόλο στη διάσκεψη της Αντίσα Μπέμπα. αλλά και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και να τηρήσουμε τις αξίες που πρεσβεύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους εσάς, τους συναδέλφους, τους παρευρισκόμενους και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ πολύ.